κλείσουμε. Item number one. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης είναι το σημείο 1. Υπάρχουν κάποιες ε, αλλαγές στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 26 θα το εξετάσουμε μετά το σημείο 8, το σημείο 31, μετά το σημείο 12 και το σημείο 10 αναβάλλεται. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι από ό,τι βλέπω. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερησία διάταξη. Περνάμε στις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Σημείο 2. Θα ήθελα να σας καλέσω σε ένα κοκτέιλ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6.30 το απόγευμα, στον Πρεσερή, είναι στο Γιάν, στον τρίτο όροφο, οργανώνεται αυτή η εκδήλωση μαζί με το Ινστιτούτο, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εμπειρογνωμοσύνης και Εμπειρογνωμόνων, που συνεδριάζει οι δικαστικοί εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη και θα παρουσιάσει ε, θα παρουσιαστεί στο κοκτέιλ το ε, νέο βιβλίο για την δικαστική εμπειρογνωμοσύνη στην Ευρώπη. Αν υπομονώ να σας καλωσορίσω μαζί με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου. Αυτά για τις ανακοινώσεις. Το σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι τα τέλη αυτής της συνεδρίασης, σε ό,τι αφορά στα πρακτικά της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Περνάμε στο σημείο 4. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Νομική Ιστορία. Να καλωσορίσουμε τους ακόλουθους εμπειρογνώμενες το δόκτωρα Μίχαλ Γκάλεντεκ από το Πανεπιστήμιο του Γκτάνσκ. Το δόκτωρα Μάθιου Ντάισον από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τον καθηγητή Dirk Χάιρμπαουτ από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης. Συγγνώμη για το προφορά μου. Και την ε, δόκτωρα Άννα Κλίματσεύσκα από το Πανεπιστήμιο του Γκτάνσκ. Uh, Αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω με ποια σειρά σκοπεύετε να πάρετε το λόγο. Όμως έχουμε στη διάθεσή μας λιγότερο από μισή ώρα. Παρακαλώ, σας δίνω το λόγο. Μπορεί η σύγκριση της νομικής ιστορίας να κατανοήσουμε τον νόμο, και να δούμε σε ποια κοινωνία βρισκόμαστε και θέλουμε να είμαστε. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία ε, σας ευχαριστεί για την δυνατότητα που μας δίνετε να απευθυνθούμε στην Επιτροπή σας ε, για το έργο μας. Ε, λέγομαι Μάθου Τάισεν και είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ισοκφόρδης και αντιπρόεδρος της εταιρείας συνάδελφος Άννα Κλιματσεύσκα, είναι επίσης ε, καθηγήτρια που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Ντάνσκ και ε, ο Τέρκ ε, Χεραμπάουτ είναι καθηγητής νομικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της γάντης και συνειδητής της εταιρείας. Έχω λάβει και έχω δώσει αρκετές διαλέξεις ε, για να ξέρω ότι ίσως να μην διασκεδάζει κανείς, ε, αν και πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο και να σας δώσω μια επισκόπηση για το ποια δουλειά κάνει η εταιρεία και τις ιδέες που παράγει. Και αν έχετε ερωτήσεις, ευχαριστώ να απαντήσουμε. Η συγκριτική νομική ιστορία μπορεί να είναι ευρεία και βαθιά όσο απαιτούν τα ερευνητικά ερωτήματα και επιτρέπει η χρηματοδότηση. Έχουμε 150 έγγραφα βάσει των οποίων μπορείτε να δείτε παραδείγματα του έργου της εταιρείας. Για πώς συνδέεται με τη δουλειά της Επιτροπής σας δρούμε σε μικρό επίπεδο και ερευνούμε στενά ερωτήματα νομικής φύσεως που αφορούν τις αποφάσεις, ε, τα άρθρα, τους ε, νομικούς πρωταγωνιστές. Μπορεί να αναφέρονται σε συγκεκριμένες μελέτες με τις οποίες ασχολείται η Επιτροπή. Παραδείγματα, πώς ε, άλλαξε η Ισπανική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Πριν ε, κάποιες δεκαετίες ε, έχουμε μια ιστορία που αφορά το γερμανικό δίκαιο και τον καθηγητή Αλμπεργούντε του Πανεπιστημίου της Τερώνα. Και η ιστορία μας δείχνει την αλληλεπίδραση μεταξύ ακαδημαϊκών και δικαστικών και πώς υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες για ε, να υπάρχει νομική μεταμόσχευση. Επίσης, είχαμε την περίπτωση που παρουσιάστηκε από το δικαστή Τζον Κόρους. Δεν ξέρω πόσο ξέρετε για το λιπεφιντορούμε, αλλά είχαμε ε, ουσιαστικά ένα εθνικό δίκαιο που ουσιαστικά εντάχθη στο ρωμαϊκό δίκαιο ε, που υπερισχύει στην Ήπειρό μας. Έχουμε ε, ουσιαστικά το θέμα της κατοχής και μπορούμε να δούμε πώς κατανοούμε αυτό τον όρο σήμερα. Το, η έννοια της κατοχής του possession είναι κάτι που συζητάμε εδώ και εκατοντάδες χρόνια και μπορούμε ίσως να μάθουμε το πώς το εθνικό δίκαιο εντάχθηκε στο ρωμαϊκό δίκαιο. Άλλα παραδείγματα αφορούν πώς ε, ο βελγικός ποινικός δόγεκα ε, το 1860 και ο Ιταλικός ποινικό ε, κώδικας δημιουργήθηκαν και επίσης ε, πώς παραδείγματος χάρη συστάθηκε και ο κώδικας για τα αυτοκίνητα και επίσης πώς παραδείγματος χάρη είχαμε ανάπτυξη του άδικου πλεονεκτήματος στο ελβετικό δίκαιο. Τώρα στο μακροεπίπεδο προσπαθούμε εδώ να κατανοήσουμε πώς αλλάζει το δίκαιο και τι σημαίνει η εθνική ταυτότητα εντός του δικαίου το πώς να κατανοήσουμε πώς ε, λαμβάνει ε, χώρα ο σχηματισμός του δικαίου μας βοηθά στο να δούμε ποιοι κανόνες έχουν εφαρμοστεί διασυνοριακά στο παρελθόν. Έχει νόημα να έχουμε ε, κανόνες που είναι ίδιοι αν ερμηνεύονται διαφορετικά στους διάφορους πολιτισμούς μπορούμε να βλέπουμε ότι είναι ίδιος τυπικά ο νόμος αλλά πρακτικά εφαρμόζεται διαφορετικά. Βέβαια υπάρχουν κάποιες δυνάμεις ε, συγκεντρωτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά και τα δύο αυτά όργανα απαιτούν διαφορετικά ειδικού παράγοντες πυροδότησης για να μπορέσουν να δράσουν ενωπημένα το δικαστήριο. Θέλει απόφαση ενό άλλου δικαστηρίου από ένα κράτο μέλο, ενώ η Κομισιόν τυπικά θα απαιτήσει κάποια κυβερνητική δράση ή αδράνεια της κυβέρνησης και ε, το μεγαλύτερο μέρος του δικαίου δεν γίνεται από τις κυβερνήσεις και δικαστικές αποφάσεις αλλά από τις δραστηριότητες των ανθρώπων και των δικηγόρων επιτόπου, των νομικών, οι οποίοι βλέπουν πώς λειτουργεί το δίκαιο. Οι περισσότεροι από την ισχύ του νόμου την ε, αισθανόμαστε χωρίς να υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου το έργο της εταιρεία ε, πολλές φορές σχηματίζει αυτή την ε, μακροεικόνα από πολλές μικρές ιστορίες που ανέφερα και άλλες φορές ξεκινά από το επίπεδο της εταιρεία και προσπαθεί να οικοδομήσει παραδείγματα. Δύο πρόσφατα παραδείγματα ε, έχουμε το έργο της, Καθηγήτρια Πιλαϊμάκη στη Φιλανδία που εξηγεί το πώς η κωδικοποίηση ε, συνεισφέρει στον εξυγχρονισμό. Οι κώδικες ε, ουσιαστικά έχουν ε, μια ζωή 200 ετών περίπου και ουσιαστικά αποτελούν παραδείγματα του τι εννοούσαμε ένα σύγχρονο νομικό σύστημα. Ίσως και αντίθετα, ο καθηγητής Μάρτιν Μπέλο από τη Σόφια έχει κάνει πολλή δουλειά για την ιδέα της Ευρώπης ως ένα παράγοντα για την οικοδόμηση μιας βουλγαρικής εθνικής ταυτότητας. Έχουμε μια αντίθετη εικόνα διαφορετικά ότι μια εθνική ταυτότητα, μια υπερεθνική ταυτότητα συνεισφέρει στην οικοδόμηση μιας εθνικής ταυτότητας. Επίσης έχουμε και παραδείγματα πώς αναπτύχθηκε η ρουμανική εθνική ταυτότητα και τα αποτελέσματα του νόμου ή της έλλειψής του στις κοινωνίες. Έχουμε και δύο συγκεκριμένα paper που αφορούσαν την πνευματική ιδιοκτησία στο ψηφιακό περιβάλλον στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ευρώπη και ιδιοτησία ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών στην πολωνική ιστορία και σε συγκριτική μελέτη με άλλες χώρες. Ένα από τα διδάγματα που προκύπτουν είναι ότι η συγκρατικό δίκαιο και η νομική ιστορία μπορούν να αποτρέψουν τρία πράγματα ότι οι κοινοί κανόνες προκύπτουν από κοινέ ανάγκες ε, σε διάφορες δικαιοδοσίες, ότι ε, κάποιοι κοινοί κανόνες έχουν ε, υιοθετηθεί μόνο αξιοκρατικά και όχι ως αποτέλεσμα ιστορικών παραγόντων και ότι ότι ε, ο νόμος που έχει ανθίσει σε ένα μόνο τόπο μπορεί να εξηγηθεί από παράγοντες που αναπτύχθηκαν μόνο σε αυτό το τόπο. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατανόηση για να βελτιώσουμε την κατάσταση του δικαίου και το πώς κατανοούμε τις κοινωνίες. Σίγουρα χρειαζόμαστε χρόνο για τη δουλειά μας, καθώς ε, για την έρευνα αυτή χρειαζόμαστε μήνες, κάνουμε έρευνα σε πολλές γλώσσες και έχουμε να κάνουμε και με διάφορα νομικό συστήματα. Το Ινστιτούτο είναι μια εταιρεία λόγιων και ερευνητών με βάση την Ευρώπη, αλλά έχουμε μέλη σε κάθε κατοικημένη γεωγραφική περιοχή και ε, ουσιαστικά κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, ε, έχουμε μέλη, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές σε όλη την Ευρώπη. Ε, πέρα από τις μεμονωμένες δημοσιεύσεις ε, έχουμε και τη δική μας εφημερίδα και φυσικά ο τίτλος είναι «Συγκριτική νομική ιστορία». Αν θέλετε έχω και κάποια αντίτυπα εδώ και ουσιαστικά ε, έχουμε σε αυτό το έγγραφο ε, πάρα πολλές μελέτες συγκριτικές στην Βαλένσια το 2010, στο Άρστερνταμ το 2012, στην Ιταλία το 2014 και στο Γκτάσκ το 2016 έχουμε οργανώσει συνεδριάσεις και οργανώνουμε και μία στο Παρίσι το 2018. Ο στόχος μας είναι να κατανοήσουμε περαιτέρω τις νομικές ιδέες πέρα από τα εθνικά σύνορα, τα εθνικά σύνορα που έχουμε σήμερα ή τα μελλοντικά. Τώρα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Άννα, ουσιαστικά για ένα ε, διάλειμμα και κατόπιν θα πάρει το λόγο και ο επόμενος συνάδελφος. Ευχαριστώ, Μάτ. Η συγκριτική νομική ιστορία μπορεί να μας ε, βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς ε, με επιτυχία μπορούμε να επιφέρουμε τη νομική αλλαγή. Το γενικότερο μήνυμα είναι ότι το περιεχόμενο ενός νομικού συστήματος και ε, η νομική κουλτούρα μπορούν να αλλάξουν με τον καιρό. Και η συγκριτική νομική ιστορία μπορεί να μας δείξει πώς ακριβώς ε, επήλθε αυτή η αλλαγή. Το 19ο αιώνα, στις αρχές του, πολυάριθμοι θεσμοί και κανόνες ε, του αυστριακού, προσικού, και αυστριακού δικαίου στις ε, πολωνικές, από τις πολωνικές αρχές και στην πολωνική επικράτεια θεωρούνταν ως ε, κάτι εξωτερικό, εξωγενές και επιβεβλημένο. Και έτσι υπήρχε αντίσταση απέναντί τους. Όμως μετά από 100 χρόνια και πάνω, κατά τη διάρκεια της ε, κωδικοποίησης και ενιαιοποίησης, διαπιστώθηκε ότι οι εκπρόσωποι επιμέρους περιφερειών ε, έδειχναν ιδιαίτερη αφοσίωση στα τοπικά τους νομικά συστήματα. Άρχισαν λοιπόν να τα περασπίζονται και πρότειναν οι διατάξεις τους να τεθούν σε ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια της ανεξάρτητης χώρας. Συχνά μάλιστα τόνιζαν ότι οι μεμονωμένες νομικές κουλτούρες είχαν απορροφηθεί από ολόκληρες γενιές νομικών, εισαγγελέων, δικαστών, ε, που τις είχαν υιοθετήσει όπως και ολόκληρη κοινωνία. Κάτι το οποίο αρχικά είχε θεωρηθεί ως εξωγενές ε, και επιβλημένο, άρχισε ο κόσμος να το υιοθετεί ως εθνική νομική του παράδοση. Αυτή η διαδικασία βέβαια πήρε καιρό. Όλοι αυτοί οι κανόνες και νόμοι έπρεπε να έχουν να υπησέλθουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ε, το νομικό και στηρίζεται από την ύπαρξη συνεκτικών και αποτελεσματικών κανόνων. Αυτή η σωστή εξίσωση για ε, την απορρόφηση εξαρτάται από τους ε, κανόνες και από το συγκείμενο, αλλά και από τις περιστάσεις. Κάποιες φορές μπορεί κάτι εξωγενές να ε, απορριφθεί κάποια στιγμή. Ενδεχομένως, το νομικό σύστημα να μην τοποθετεί σωστά την προέλευση αυτού του ξένου στοιχείου. Το πλέον σύνηθε στερεότυπο, για παράδειγμα, για το πολωνικό εμπορικό δίκαιο είναι ότι οι ισχύοντε κανόνε βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στο γερμανικό εμπορικό δίκαιο του 1897. Ταυτόχρονα, το πολωνικό εμπορικό δίκαιο προέκυψε στην, στο μεσοδιάστημα μετά την ε, έκδοση αυτού του ε, εμπορικού δικαίου. Πολλοί σχολιαστές εκείνη την περίοδο προσπάθησαν να ε, δείξουν ότι ποια ήταν η πηγή συγκεκριμένων διατάξεων, συγκρίνοντας τα μόνο κυριολεκτικά με το περιεχόμενο άλλων ευρωπαϊκών κωδίκων, πιο συγκεκριμένα με το γερμανικό εμπορικό δίκαιο του 1897. Όμως, σε μεγάλο βαθμό ξεχνάμε σήμερα ότι σε μεγάλο βαθμό το υπόβαθρο του πολωνικού εμπορικού δικαίου προήλθε από την γαλλική νομική κουλτούρα. Αυτή είναι η συνταγματική και νομοθετική βάση, δηλαδή, που προέκυψε από το γαλλικό δίκαιο. Διατάξεις του γαλλικού εμπορικού δικαίου ίσχυσαν στην Πολωνία για πάνω από έναν αιώνα και ολόκληρες γενναίες νομικών και δικαστών τις απορρόφησαν. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι οι συντάκτες του Γενικού Γερμανικού ε, Εμπορικού Κώδικα του 1861 πριν δηλαδή το 1897, σε μεγάλο βαθμό βασίστηκαν στις, γερμα... στις, της στις γαλλικές διατάξεις. Επομένως, το υπόβαθρο για το γερμανικό μοντέλο εμπορικού δικαίου δεν δημιουργήθηκε εν κενό. Η νομική μας ιστορία, λοιπόν, είναι πολύ περισσότερο διασυνδεδεμένη από ό,τι συνειδητοποιούμε. Σε αυτή τη διαδικασία απορρόφησης ή υιοθέτηση με την πάρτα του καιρού, μπορούμε να αναφερθούμε ε, στα αξιοκρατικά κριτήρια. Υπάρχουν ορισμένα ιδεολογικά κριτήρια τα οποία γίνονται δεκτά από μία κοινωνία και έχουν εγγραφεί ε, στην ε, κουλτούρα μιας χώρας. Είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα κανείς να απαλείψει. Το 19ο αιώνα λοιπόν υπήρξε μια μακροσκελής ε, και έντονη συζήτηση σχετικά με την ε, παρέκκληση από τον ε, γαλλικό αστικό κώδικα που μεταξύ άλλων είχε εισαγάγει και τον θεσμό του πολιτικού γάμου. Τα πράγματα κάπως ηρέμησαν μετά την αναθεώρηση αυτών των διατάξεων όταν επανεκδηθήθηκε η, ε, ο θρησκευτικό γάμος. Έτσι, επεβίωσε αυτός ο κώδικας στην Πολωνία μέχρι το 1946. Οι πρόσφατες αντιδράσεις κατά της, ε, του περιορισμού, ε, της θέσπισης περιορισμών στο νόμο περί αμβλώσεων στην Πολωνία είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνει πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε ε, το δίκαιο με κάποιες επεπιθήσεις ε, λαϊκές, αν θέλετε. Γι' αυτό δεν είναι το πλέον σημαντικό να θεσπίζονται ε, νομικές διατάξεις από τις εθνικές νομικές αρχές. Ευχαριστώ. Όπως ακούσατε από του συναδέλφου, ένα από του στόχου τη κοινωνία μας είναι να εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι να έχουν συνείδηση των εθνικών ε, παραδόσεων στην Ευρώπη και ε, στηρίζονται σε μια γόνιμη ανταλλαγή ιδεών. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει ένα εργαστήριο παραγωγή δικαίου. Ωστόσο, η συγκριτική ιστορία μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το πώς νέοι κανόνες ή νέα θεσμικά όργανα μπορούν να διαδραματίσουν ε, καθοριστικό ρόλο στον πραγματικό κόσμο όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Στην κοινωνία μας θέλουμε να ανοίξουμε ε, να συγκεντρώσουμε τις ιδέες όχι μόνο από μία χώρα και τα μέλη της, αλλά από όλες τις χώρες. Και θα ήθελα να σας ε, δώσω ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι, αναφέρονται, ε, επιθυμούν έναν ενιαίο αστικό κώδικα για την Ευρώπη. Ορισμένοι ε, συμφωνούν, άλλοι το θεωρούν εφιάλτη, άλλοι εφικτή πραγματικότητα, άλλοι μια παράλογη ιδέα, αλλά μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για κάτι καινοφανές. Άρα μιλάμε χωρίς να στεριζόμαστε στα πραγματικά δεδομένα. Ωστόσο η συγκριτική νομική ιστορία μπορεί να μας δώσει μια δυνατότητα σύγκρισης η ενοποίηση του δικαίου στο Γερμανία έγινε το 19ο αιώνα. Και υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί γιατί υπήρχαν πολλά κρατήδια στη Γερμανία τότε και τώρα υπάρχουν πολλά κράτη στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μπορεί να συγκριθεί με το γερμανικό Reichstag ε, η Επιτροπή με το Reichsamt το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με το υψηλό δικαστήριο το Reichsgericht και ούτω καθεξής. Ωστόσο, δεν είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστούν και διαφορές. Για παράδειγμα, ε, το αίτημα ενιαίου κώδικα ε, δεν ε, είναι τόσο αισθητό σήμερα στην Ευρώπη όσο στο παρελθόν στη Γερμανία. Ωστόσο, στη Γερμανία, της εποχής εκείνης ριζώνει η ιδέα ότι χρειάζεται ένα νέο γερμανικό δίκαιο και ε, όπως η Γερμανία της εποχής εκείνης η Ευρώπη δεν έχει μία μόνο γλώσσα και ούτε έχει και νέο πολιτισμό και Άρα μπορεί κανείς να αμφιβάλλει για το κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρχει ένας ενιαίος ε, νομικός ε, κώδικας για όλη την Ευρώπη. Ωστόσο η γερμανική ιστορία δείχνει ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα σε λιγότερο από ένα αιώνα. Και το 1840 υπήρξε το αίτημα ενός ενιαίου νομικού συστήματος στη Γερμανία. Και άμεσα αυτό, ε, αμφισβητήθηκε αλλά στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένας ενιαίος κώδικας και αυτό δείχνει ότι παρά τις διαφορές υπάρχουν πολλοί ενδυνάμοι παραλληλισμοί ε, μεταξύ των ε, παραγόντων που ήταν υπέρ της ενοποίησης του ιδιωτικού δικαίου το 19ο αιώνα στη Γερμανία και αυτού που διαδραματίζεται σήμερα στην Ευρώπη. Η στάση των πολιτών είναι παραπλήσια και υπάρχει μια, γιατί υπάρχει μια παρουσία κοινών πολιτικών θεσμικών οργάνων και δικαστηρίων σε υψηλό βαθμό ε, μιας γραφειοκρατίας και υπάρχει μια νέα ιδεολογία των δικαιοδοτικών συστημάτων τα οποία ενέχονται εδώ. Και δεδομένων όλων αυτών των ε, ομοιοτήτων δικαιολογείται το ερώτημα κατά πόσο το παρελθόν της Γερμανίας ε, μπορεί να μας δώσει κάποια διδάγματα για, τα μελλοντικά, για το μελλοντικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών ε, συστημάτων αστικού δικαίου. Έχω φέρει κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να σας παρουσιάσω για παράδειγμα ότι βεβαίως το δίκαιο αυτό δεν μπορεί να συνταχθεί από ένα μόνο πρόσωπο, αλλά από μια επιτροπή ή από μια τριμελή επιτροπή νομικών εμπειρογνωμόνων και μια επιτροπή πολιτικών εκπροσώπων και ομάδων ε, κοινωνικών συμφερόντων. Επίσης, ένας τέτοιος κώδικας χρειάζεται, ένα ψηλό, ε, ε, χρειάζεται μια διαθεση σε ανώτατο επίπεδο και ε, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο προσαρμογής, ερμηνείας και εξέλιξης του δικαίου. Ένα σχέδιο νομικού συστήματος δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπερβολικά ε, μακροσκελείς και σύνθετες συζητήσεις όπως ο γάμος μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου. Τώρα, αυτά είναι κάποια, κάποιες γενικές σκέψεις, το γενικό πλαίσιο. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ την προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι πριν καταλήξουμε σε ένα τέτοιο τεράστιο εγχείρημα, όπως είναι ένα κοινό σχέδιο αστικού κώδικα για ολόκληρη την Ευρώπη, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ενιαία, ένα ενιαίο νομικό πολιτισμό. Και τώρα στην ευρωπαϊκή κοινωνία γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να διαμορφωθεί μια ενιαία, ένας ενιαίος νομικός πολιτισμός, το οποίο δεν θα είναι μια μόνο καλλιέργεια, μια μονοκουλτούρα, αλλά θα υπάρχει κάτι το οποίο θα γεφυρώνει τη γερμανική νομική ιστορία, ε, παράλληλα με την ιστορία της ε, Γαλλίας, και της ε, Πολωνίας. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη συνέχεια εναπόκειται στα χέρια των... Ε, θα συμβεί στη συνέχεια εναπόκειται στους ε, πολιτικούς. Εμείς απλώς μελετούμε την νομική ιστορία, δεν την διαμορφώνουμε, εσείς τη διαμορφώνετε. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν την ιστορία παρά, δεν τη μελετούν, αλλά δεν μελετούν το παρελθόν, αλλά ορισμένες φορές προτιμούν νέες ε, λύσεις. Γιατί η βασική ιδέα δεν είναι να αξιοποιηθεί η ιστορία επαναλαμβάνοντας την, αλλά να αξιοποιηθεί πηγαίνοντας πέρα από τα όρια της. Ε, δηλαδή βασιζόμενοι στο παρελθόν να το ξεπεράσουμε. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Δεν ξέρουμε πόσο η εταιρεία για τη συγκρίτη κοινωνική ιστορία μπορεί να βοηθήσει. Ξέρουμε τη δουλειά που κάνουμε αρχικά. Γίνεται για την ακαδημαϊκή έρευνα. Θέλουμε να ξέρουμε την αλήθεια και να μπορούμε να την αποδείξουμε. Παρ' όλα αυτά, ταυτόχρονα, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, παρακαλώ ρωτήστε, ζητήστε το μας. Uh, Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ, για τις παρουσιάσεις σας μας προσχέσατε τη σημαντική δραστηριότητά σας. Υπάρχουν ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριος Βιεύκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι ερώτηση, απλώς θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας που δέχτηκαν να παρευρεθούν εδώ. Ήθελα να πω το εξής. Εσείς με αυτή τη συγκριτική δουλειά που κάνετε θα έπρεπε να ανοίξετε τα μάτια στους νομοθέτες και σε όλους αυτούς που χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή το δίκαιο. Υπάρχουν ε, διάφορες επιρροές, αυτό το βλέπουμε εδώ και αιώνες, γιατί τι κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Προσπαθούμε να βρούμε ελάχιστους κανόνες ε, για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Πριν 200-300 χρόνια υπήρχαν κάποιες ε, εντάσεις και σήμερα υπάρχουν, όμως η δική σας δουλειά ουσιαστικά μας δείχνει μια διαφορετική σκοπιά, ότι δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε αλλά θα πρέπει να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας. Αυτό λέμε πολλές φορές, να καλλιεργήσουμε έναν ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό που να είναι κοινό, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γι' αυτό και αυτός ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός είναι που θα μας δώσει νέες δυνατότητες. Ο καθηγητής Μπέρλιγκερ το επανελάμβανε συχνά ότι δίχως ένα κοινό νομικό πολιτισμό θα είναι δύσκολο για μας στο μέλλον να πετύχουμε μια ιστορική στιγμή, δηλαδή να έχουμε μια ιστορική λύση που να αποτελεί καλό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για το πόσο καλά λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, η συνεργασία μας δεν μπορεί να βασίζεται σε πάρα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, όμως αυτή η εστίαση και το ότι βλέπουμε ότι με το πέρασμα του χρόνου αλληλοσυνδέονται διάφορα στοιχεία, ε, είναι ουσιαστικά ένας τρόπος εργασίας πάρα πολύ χρήσιμος για μας. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τις ε, παρουσιάσεις που εν μέρη άκουσα αλλά τράβηξε την προσοχή μου το εξής, κύριε Χερμπό. Είπατε ότι για να αναπτυχθεί ένας κοινό νομικός πολιτισμός στην Ευρώπη πρέπει οι άνθρωποι από διάφορες περιφέρειες και από διάφορους νομικούς πολιτισμούς να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Θα ήθελα να πω πόσο εύκολο είναι να υπάρχουν όμως κάποιες προκαταλήψεις και να ξεχάσουμε κάποιους, γιατί αναφέρεται τις μεγάλες χώρες και τις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως μπορείτε να μας πείτε τι μπορούμε να μάθουμε πιο περιφερειακές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη τις σκανδιναβικές χώρες, μήπως το ερευνήσετε αυτό. Νομίζω ότι έχετε δίκιο στην ερώτησή σας. Δηλαδή, Λέτε ότι όλοι έχουν κατά νου τις μεγάλες χώρες, αλλά και εγώ ίδιος έρχομαι από μια μικρή χώρα, από το Βέλγιο. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί ένα από τα πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε είναι να ακούσουν οι άνθρωποι για τις υπόλοιπες χώρες και να τους ενθαρρύνουμε εστιάζεται να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ε, και άλλες χώρες πέρα από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί θέλουμε ουσιαστικά να λάβουμε υπόψη και τις υπόλοιπες χώρες. Και στις συναντήσεις της εταιρεία ακριβώς αυτό συνέβαινε. Δηλαδή, να έχουμε ανθρώπους που να μας ε, κάνουν κάποιε παρουσιάσει όχι μόνο από τι σκανδιναβικέ χώρε που τι γνωρίζω πολύ καλά, γιατί έχω μεταβεί πάρα πολλέ φορέ στη Φιλανδία, στην Νορβηγία, στη Σουηδία, αλλά και από άλλε χώρε. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογή διευρύνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αρχικά είχαμε μόνο τα παραδοσιακά κρατημέλη, τα πρώτα κρατημέλη που ίδρυσαν την Ένωση. Όμως, τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διευρυνθεί και η νομική ιστορία. Και μόλις έλαβα από τους Πολωνούς φίλους μου ένα βιβλίο, το πρώτο βιβλίο για την νομική ιστορία της Πολωνίας στα αγγλικά. Υπάρχουν ε, και πολλές άλλες γνώσεις ε, που ε, μπορώ να διαβάσω. Δεν μπορούσα να διαβάσω πολωνικά, αλλά τώρα έχω το βιβλίο αυτό. Μπορείτε να το δείτε. Αυτό ακριβώς θέλουμε να ενθαρρύνουμε, να κάνουν οι άνθρωποι αυτό, όχι μόνο στα αγγλικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες, γιατί και όχι στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε λοιπόν κάτι τέτοιο για να μην έχουμε και μόνο καλλιέργεια στο επίπεδο της γλώσσας. Δηλαδή όχι μόνο μία χώρα ούτε μόνο μία γλώσσα. Γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε τώρα σας δίνει τώρα τη λάθος εντύπωση. Thank you, Ευχαριστώ κύριε monsieur. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, τους εκπροσώπους ε, της εταιρεία για την συγκριτική νομική ιστορία, ως και εγώ καθηγητής ε, δικαίου θεωρώ ότι η συγκριτική ε, νομική ιστορία είναι πολύ σημαντικό πεδίο γιατί μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την κοινή μας ιστορία και τις αλληλεπιδράσεις που είχαμε στην ευρωπαϊκή ιστορία. Για παράδειγμα, μας δώσατε ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα στην Πολωνία που άντλησε έμπνευση από το γερμανικό και γαλλικό δίκαιο. Αυτό είναι στοιχείο που ε, μας δίνει τροφή για σκέψη. Εγώ προφανώ και θέλω να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια διερεύνησης ε, της συγκριτικής νομικής ιστορίας. Για μας είναι μια πηγή προβληματισμού αυτό και συμφωνώ με τα όσο υπόθηκαν ότι θα πρέπει να ε, στηριχθούμε στο παρελθόν για να διαμορφώσουμε το μέλλον. Είναι ένα κοινό σημείο που έχουμε θεωρώ. Εκεί όμως που δεν συμφωνώ τόσο είναι όταν συγκεκριμένοι παρεμβαίνοντες μεταξύ των ευρωβουλευτών Προσπαθούν να αξιοποιήσουν ε, τη ε, συγκριτική νομική ιστορία ε, για ιδεολογικούς σκοπούς. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Είμαι υπέρ τα ευρωπαϊκά δίκαια να συνεχίσουν να εμπλουτίζουν το ένα το άλλο μέσω αμοιβαίων δανείων. Αυτό θα έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται. Όμως δεν θέλω μία ενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου γιατί ξέρουμε και τους περιορισμούς που προκύπτουν από την συγκριτική νομική ιστορία. Θέλετε να εξαλείψετε τον πλούτο ε, του ευρωπαϊκού, των ευρωπαϊκών δικαίων μάλλον με την ε, υπερβολική ενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Όπως και με τα κράτη, ε, συνεργασία, συντονισμός με στήριξη των ευρωπαϊκών δικαίων, αλλά χωρίς να υπάρχει μία και μόνο νομική τάξη. Και μάλιστα καταγγέλλω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάνει αυτή την προσπάθεια και προωθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Δίκαιο και έτσι θεωρώ ότι θέλουν ε, να θέσουν ένα τέλος στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ μορφές δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Η ενότητα αλλά και διαφοροποίηση, κύριε Λευγετών, δεν χρειάζεται να φοβάστε γιατί είναι βασικό αξίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι βέβαια να προτείνει ε, την ε, ενοποίηση. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους ε, αξιότιμους προσκεκλημένους μας για την παρουσία τους εδώ. Είναι σημαντικό που μας παρουσιάσατε το έργο σας και έτσι γνωρίζουμε την ύπαρξη της εταιρεία σας και ότι αν χρειαστεί έχουμε ένα σημαντικό εταίρο με τον οποίο μπορούμε να συνομιλήσουμε. Ευχαριστούμε. We continue Συνεχίζουμε τώρα με το σημείο 5 εξέταση τροπολογιών για την ε, διασυνοριακή φορητότητα των επιγραμμικών ε, υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Ο κύριος Ζωμαρή Καβαντά, εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την συμμετοχή τους ε, στις εργασίες για αυτή την εισήγηση και την επικοδομητική συμβολή τους στις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει ε, και μέχρι το τέλος την ψηφοφορία στο πλαίσιο της Επιτροπής Γιούρη σε μερικές εβδομάδες έχουμε εξετάσει το σύνολο των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί για την ε, πρόταση κανονισμού της Επιτροπής και βλέπουμε ότι το σύνολο των ε, σημείων που αφορούν αυτό το φάκελο μπορούν να αποτελούσουν αντικείμενο συνένεσης, όχι μόνο στο πλαίσιο της Επιτροπής Γιούρη, αυτό δεν θα είναι δύσκολο εξάλλου πιστεύω, αλλά και στην ε, καθήλυνα αρμόδια που είναι η Επιτροπή ε, Πολιτισμού ΙΜΚΟ και ΙΤΡΕ. Επομένω, ε, θα ήθελα με, τη, με το μεγαλύτερο δυνατό συμβασμό να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση για αυτό το φάκελο και ε, είμαστε στη διάθεσή σας. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Πριν περάσω στην ουσία, θα ήθελα να σας αναφέρω το χρονοδιάγραμμα που προτείνουμε. 20 Οκτωβρίου θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση των σκιωδών για ε, την ε, πρόταση αυτή. 20 Οκτωβρίου. 8 Νοεμβρίου υπάρχει δυνατότητα δεύτερη συνάντηση σκιωδών. Μεταξύ των δύο συναντήσεων, μεταξύ 20 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρίου δηλαδή, οι ομάδες μας θα εργαστούν από κοινού ε, για να επεξεργαστούν ε, πιθανές ε, συμβαστικές τροπολογίες. Και 28 Νοεμβρίου θα ψηφιστεί η έκθεση στην Επιτροπή Γιούρη. 20 Οκτωβρίου λοιπόν αρχικά, μετά 8 Νοεμβρίου και 28 Νοεμβρίου τέλος. Τώρα, ας περάσουμε στην ουσία. για τις διαπραγματεύσεις. Βάσει των επιμέρους τροπολογιών της Γιούρη και των γνωμοδοτήσεων των ε, επιμέρους επιτροπών, βλέπουμε ότι οι συστάσεις που θα προτείνω ε, στους εστιώδεις είναι οι εξή. Πρώτον, στο πλαίσιο του κανονισμού θέλουμε ε, να διασφαλίσουμε ότι η φορητότητα επιτρέπει σε έναν συνδρομητή να έχει πρόσβαση ε, στις υπηρεσίες που έχει ε, αγοράσει, ακόμα και όταν μεταβαίνει σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, πρώτερη ταυτοποίηση του κράτους μέλους διαμονής του, προφανώς. Δεύτερον, στήριξη των δικαιωμάτων γενετικής ιδιοκτησίας και αυτά θα πρέπει να διασφαλίζονται μέσω του παρόχου. Τρίτον, ε, ε μη επιβολή επιπλέον κόστους ή χρέωσης για την φορητότητα. Η διασυνοριακή φορητότητα λοιπόν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξομοιώνεται με την διασυνοριακή πρόσβαση Βεβαίω με την επιφύλαξη των ε, επιπέδων προστασίας ε, που έχουν ήδη θεσπιστεί, Εμεί δεν θέλουμε να αποσυντονίσουμε και να αποσταθεροποιήσουμε ε, τις αγορές και πιο συγκεκριμένα την αγορά καλλιτεχνική δημιουργία. Ως προς τον ορισμό της προσωρινή παρουσίας του συνδρομητή εκτός της χώρας διαμονής του και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να, στο οποίο θα πρέπει να καταλήξουμε. Από ό,τι φαίνεται όλοι συμφωνούν να πούμε ότι, υπάρχει, ε, ότι πρόκειται για μια προσωρινή περίοδο εκτός του κράτους μέλους ε, όπου διαμένει ε, μόνιμα ο συνδρομητής. Σκόπιμο θα ήταν να προσδιορίσουμε ότι η περίοδος αυτή που περνάει ο συνδρομητής σε άλλη χώρα δεν θα πρέπει να είναι περιορισμένη στον χρόνο, να μην ορίζεται δηλαδή, γιατί είναι ιδιαίτερα σύνθετο για τον ορισμό των επιγραμμικών ε, υπηρεσιών ή υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου. Εδώ πρέπει να υπάρχει για όλες τις ε, δωρεάν υπηρεσίες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Και βλέπω με χαρά ότι ε, συμφωνούμε όλοι σε αυτή την πρόταση για τους παρόχους ε, υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου που έχουν ε, ε, τοπικές υποδομές. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πρόβλημα να δίνουν πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο υπό συγκεκριμένη αδειοδότηση επιπλέον του περιεχομένου το οποίο, στο οποίο έχει πρόσβαση στη χώρα διαμονής του. Μετά, κάτι ακόμα ε, για, τον, ε, για την ειλικρίνεια του συνδρομητή. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της φορητότητας. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι η δήλωση ε, τόπου διαμονής είναι ειλικρινής και επαληθεύσιμη. Τώρα, τρία συμπεράσματα είναι, έχουμε βασικά. Πρώτον, ε, δήλωση λόγω τιμής ε, μετά δεν θα πρέπει να ζητούμε από τον συνδρομητή να προσκομίσει πάνω από δύο μέσα επαλήθευσης. Δεν θέλουμε κι εμείς ε, να λειτουργήσουμε ως αστυνομικές αρχές για τους συνδρομητές. Μετά σε περίπτωση σκο... εύλογης μάλλον φιβολίας, θα πρέπει ο πάροχος να ε, ε, δύναται να ζητήσει από τον συνδρομητή και πάλι να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία για την απαλήθευση του κράτους μέλους διαμονής του. Ε, δεν είναι κάτι το τρομερό, αλλά είναι μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας. Ότι και ο συνδρομητής και ο πάροχος τηρούν τις του όρου που έχουμε θεσπίσει. Μένω στη διάθεσή σα, για περαιτέρω πληροφορίες και για περαιτέρω συζητήσει για την έκθεση αυτή. Τώρα, για την απαγόρευση συγκεκριμένων ε, συμβατικών ρητρών για τον περιορισμό της φορητότητα. Η φορητότητα δεν θα πρέπει να περιορίζεται, κατά τη γνώμη μου, από καμία ε, συμβατική ρήτρα, εκτός από μία. Αυτή που επιτρέπει στον πάροχο να μην προσφέρει τη φορητότητα στον συνδρομητή που δεν έχει προσκομίσει το ή τα απαραίτητα έγγραφα για την επαλήθευση της ε, ε δήλωσής του για το κράτος μέλος διαμονής του. Σε ό,τι αφορά την ε, αξιολόγηση αντικτύπου μετά από τρία χρόνια θέση σε σχέση του κανονισμού. Είμαι υπέρ μια τέτοια ε, αξιολόγηση αντικτύπου προκειμένου να αξιολογήσουμε και την αποτελεσματικότητα των μέσων επαλήθευσης που έχουμε ε, επιλέξει και για να εντοπίσουμε τυχόν εξελίξεις στον κλάδο που μπορεί να έχουν ανακύψει ε, μέσα στην τριετία. Γιατί ξέρουμε ότι όλα αυτά που άπτονται των οπτικοακουστικών, ε, του περιεχομένου κτλ. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα κινούνται πολύ γρήγορα. Δεν πρέπει να ε, κλειστούμε και να περιοριστούμε σε έναν κανονισμό. Να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα αναθεώρησης στη συνέχεια. Μετά, θέση σε ισχύ εντός 12 μηνών θεωρώ και τίποτα δεν εμποδίζει τους ε, παρόχους υπηρεσιών να θέσουν σε ισχύ τη φορητότητα των υπηρεσιών τους και πιο πριν γιατί όπως και να έχει θα γίνει. Ας έχουν λοιπόν και την δυνατότητα να κινηθούν πιο γρήγορα οι πάροχοι. Αυτά θέλω να θέσω υπό την προσοχή σας, ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκο Τσούλο από την ΙΜΚΟ και γιατί όπως γνωρίζετε η ΙΜΚΟ ε, βάσει του κανόνα 54 συνδέεται στην σύνταξη, συμμετέχει στη σύνταξη. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μπορώ να παρέμβω για το έγγραφο που εγκρίθηκε στην ΙΜΚΟ σε αυτή την επιτροφή. Κατανοώ ε, τους λόγους ε, που σας όθησαν να συμμετέχετε στην ψηφοφορία και εμείς συνειδητοποίησαμε ότι πρόκειται για μια πιο πολύπλοκη έκθεση από ό,τι μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Πρέπει όμως να πω ότι εμείς είχαμε δεκτεί για κάποιες πιέσεις ε, για να μπορούμε να έχουμε έτοιμη την έκθεση για να τη λάβετε εγκαίρως και πολλές φορές υπογραμμίζεται ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και δυστυχώς ε, βλέπουμε ε, ότι υπήρχε μια κάποια καθυστερήση, όμως ε, τελικά φτάσαμε σε ένα στο κείμενο με το οποίο πολλοί συμφωνούν. Η ΚΟ για όλο το κείμενο γνωμοδότησε δυνάμει του άρθρου 54 και ασχοληθήκαμε με όλα τα άρθρα και σχεδόν ομόφωνα εγκρίθηκε το κείμενο 33 ψήφοι υπέρ στις 34 και είχαμε τη συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων της Επιτροπής ε, και εδώ περιλαμβάνονται πολλές αρχές οι οποίες είναι σημαντικές για την ΙΜΚΟ και μπορώ να πω ότι ε, ο κύριος Καβαντά από ό,τι φαίνεται συμφωνεί σε πολλά σημεία και αυτό με ικανοποιεί. Παραδείγματος χάρη προκύπτει η βούληση να υπάρχει διαφοροποίηση τη φορετότητας ε, από την ε, διασυνοριακή πρόσβαση χωρίς διακρίσεις. Επικεντρωθήκαμε στα δικαιώματα και τις ευκαιρίες για τον καταναλωτή, αλλά θέλουμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχει και υπερβολικό άχθος. Γι' αυτό ως ε, μέσα επαλήθευσης είπαμε ότι ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά παραβίαση του απορρίτου αλλά τα μέρη της επαλήθευσης θα πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν τη σωστή λειτουργία του συστήματος φορητότητας. Αυτό το λέμε και από την αρχή και στο κείμενο προκύπτει γιατί είναι η καρδιά της λειτουργίας του. ησυχήσαμε, θέλαμε να τονίσουμε ότι το θέμα της φορητότητας δεν θα πρέπει να αλλάξει τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στο κλάδο και ε, επίσης θέλαμε να υπάρχει απαραίτητη ποιότητα της υπηρεσίας. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό αν δεν δίναμε και τις απαραίτητες πληροφορίες στον καταναλωτή. Επίσης είπαμε σαφήνεια ότι δεν είναι δυνατό ε, να καταστραγηθεί ο κανονισμός εφαρμόζοντας τον κανόνα μιας τρίτης χώρας. Επίσης είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι παίρνουμε μια θέση ισχυρή υπέρ του καταναλωτή και προστατεύουμε τον κλάδο και το μοντέλο χρηματοδότησής του. Έτσι λοιπόν το κείμενο του κυρίου Καβαντά ήδη έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με το δικό μας και αποτελεί εξαιρετική βάση. Ξεκινάμε από κοντινές θέσεις και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα τελικό κείμενο που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων επιτροπών και να έχουμε μια ισχυρή θέση ως Κοινοβούλιο τη στιγμή που θα έρθουμε να διαπραγματευτούμε το Συμβούλιο. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η κυρία Σαμπίνε Φερχάιεν από την Επιτροπή Πολιτισμού βάσει επίσης του άρθρου 54 συντάκτρια. Ναι, καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Καβαντά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού μπορούμε να δώσουμε τη δική μας γνωμοδότηση και να επισημάνουμε τα σημαντικά στοιχεία στην επί της αρμόδια ε, Επιτροπή. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζουμε πάρα πολύ το γεγονός ότι στους ε, βασικούς μας προσανατολισμούς όσον αφορά ε, το σχέδιο έκθεσης δεν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις όσον αφορά τις βασικές προθέσεις σε σχέση με μια φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, κυρίως των οπτικοακουστικών περιεχομένων. Για μας ήταν σημαντικό να γίνει σεβαστή η αρχή της εδαφικότητας, καθώς και η αρχή μιας επαρκούς προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων τα οποία πραγματικά να είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες, ούτως ώστε να υπάρξει πράγματι μία φορητότητα και όχι μία, να εξασφαλιστεί μία προσβασιμότητα από την πίσω πόρτα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η άποψη και πραγματικά υιοθετήθηκε από την Νομική Επιτροπή. Ε, εδώ η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ε, δεν ε, διατυπώνει ε, χρονικές προθεσμίες και αυτό ήταν σημαντικό στο πλαίσιο της συζήτησης για να μην υπάρχει και πάλι συγκαλυμμένη προσβασιμότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για αυτή την γενναιόδορη πρόταση όσον αφορά τα, τις χρονικές, τους χρονικούς περιορισμούς. Ε, εδώ είναι πολύ σημαντικό και αυτό το καθιστάμε σαφέ στην Επιτροπή Πολιτισμού να καταλήξουμε σε σωστού ορισμού. Γι' αυτό χαιρετίζουμε το γεγονό ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στηρίχθηκε σε δύο κριτήρια τα οποία θα πρέπει να υιοθετηθούν όσον αφορά ε, τον έλεγχο, τη διενέργεια των ελέγχων. Και εμεί είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε δύο κριτήρια, αλλά όχι ε, περισσότερα, γιατί υπάρχουν και κάποια πιο αδύναμα κριτήρια όσον αφορά τον έλεγχο του τόπου κατοικίας. Γι' αυτό θα έπρεπε να σταθμίσουμε πραγματικά ποια είναι τα κατάλληλα κριτήρια και ποια όχι. Ε, γι' αυτό είπαμε ότι δύο είναι καλός ε, αριθμός, τουλάχιστον δύο. Τώρα, όσον αφορά την αρχή της δαφικότητας, ε, την θέσαμε στο κέντρο της προσοχής μας γιατί είναι σημαντικό όσον αφορά την τήρηση της πολυμορφίας στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και τα μοντέλα χρηματοδότησης καθώς και η βάση της χρηματοδότησης πολυμορφίας εξαρτάται από την εδαφική ε, αδειοδότηση. Ε, ε, και δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μια ομογενοποίηση όσον αφορά την αδειοδότηση. Λοιπόν, υπάρχουν ε, δυνατότητες για δωρεάν υπηρεσίες όπως είναι το free to the air, να γίνουν φορητές αυτές οι υπηρεσίες ως opt-in και αυτό το είχαμε προβλέψει εμείς, να υπάρξει αυτή η δυνατότητα για παρόχους περιεχομένων ή παρόχους υπηρεσιών που έχουν επιγραμμικές υπηρεσίες που να προσφέρονται δωρεάν. Ε, μπορεί λοιπόν να υπάρξουν ως opt-in, αλλά όχι υποχρεωτικά. Τώρα, όσον αφορά την ε, παλήθευση, ε, θεωρώ ότι πραγματικά είναι και προς συμφέρον των παρόχων να υπάρξει μία φορητότητα, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μία βελτίωση των υπηρεσιών. Και πάλι θα ήθελα να πω ότι οι απόψεις των δύο υποτερπών συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο νομοθεσίες εδώ, διαπιστώνουμε ότι ε, ε, πραγματικά θα τύχουν τις επιδοκιμασίες ε, πολλών Ευρωπαίων πολιτών ε, οι οποίοι, ε, γιατί με τον τρόπο αυτό θα λύσουν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή και θα μπορέσουν ε, να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις φορητές πλέον υπηρεσίες, τις φορητές πλέον, τα φορητά πλέον περιεχόμενα εκπομπών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο εξωτερικό για σπουδές ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αυτή τη στιγμή έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές στη χώρα διαμονής τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη ανακούφιση για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσει των ε, χρηστών, των πολιτών. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που και η, Επιτροπή της, και η, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και αυτή δεν εμφανίζει σοβαρές ε, αποκλήσεις από τη δική μας και από αυτήν της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η κυρία Αγκάτα Γέρμπα, τη Γενική Διεύθυνση Connect. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε συγκεκριμένε παρατηρήσει. Χαιρετίζουμε την ε, έκθεση του κυρίου Καβαντά. Βλέπουμε στη συνέχιση των συζητήσεων και χαιρετίζουμε το γεγονό ότι μένεται αρκετά κοντά στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι πιο σημαντικές αρχές στις οποίες ε, βασίζεται αυτή η πρόταση, η υποχρέωση δηλαδή παροχής φορητότητας, διατηρείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Κέστερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καβατά για την ε, πραγματικά αξιόλογη εργασία σας, για την ε, καλή βάση ε, που δημιουργήσατε συζήτησης πραγματικά συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και η συζήτηση έδειξε ότι υπάρχει μια συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων επί πολλών θεμάτων. Κυρίως συμφωνούμε όλοι για το γεγονός ότι οι χρήστες ε, χωρίς, ε, χρονικά, χωρίς χρονικούς προορισμούς, περιορισμούς θα πρέπει να μπορούν να υποφελούνται από την φορητότητα των υπηρεσιών χωρίς επιπλέον κόστη για τη χρήση της φορητότητας και επίσης συμφωνούμε για το γεγονός ότι οι χρήστες ε, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο τοπικό ρεπερτόριο ε, μιας επιγραμμικής υπηρεσίας όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Ένα επίμαχο σημείο είναι το θέμα του ελέγχου. Και χαίρομαι που εδώ μετα... στις προτάσεις πολλών άλλων συναδέλφων δεν ε, συμπεριλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των μέσων επαλήθευσης γιατί ένα ε, checking δεν θεωρώ ότι είναι αποτελεσματικό και είναι αφίβολο όσον αφορά ε, την επαρκή προστασία των δεδομένων. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η άποψη συμπεριλήφθη στις ε, γνωμοδοτήσεις της ΙΜΚΟ και της ΙΤΡΑ. Και ελπίζω ότι θα μπορούμε και μελλοντικά να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τους Και θα ήθελα να επισέλθω επίση σε κάποια σημεία τα οποία στι περαιτέρω διαβουλεύσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθούν. Το πρώτο αφορά τον έλεγχο της προσωρινής ε, διαμονής στη βάση αυτών των ελέγχων στις τροπολογίες 215 ε, ε, και 218 ε, απευθύνεται η σύσταση να γίνεται αυτό το beat checking, IP checking ε, και διερωτώ με ε, σε ποια βάση θα πρέπει να γίνεται αυτό το IP checking. Εάν ε, δεν βρίσκεται κάποιος σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα γίνει. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε είναι το ζήτημα της ε, οδετερότητας των τεχνολογικών μέσων. Ορισμένες τροπολογίες έχουν σαν σκοπό ε, να υποχρεώσουν τους παρόχους να, ε, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ουδέτερα ως προς τα τεχνολογικά μέσα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνει. Το τρίτο αφορά τις αρχές που θα πρέπει να διενεργήσουν τον έλεγχο Κύριε Καβαντά, θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε περαιτέρω κατά πόσο η σύσταση μιας τέτοιας ε, ελεγκτική, ε, αρχής έχει νόημα γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για την, το υπερβολικό γραφειοκρατικό άχθος και ενδεχομένως μια τέτοια αρχή τελικά δεν ξέρω κατά πόσο θα είχε νόημα. Θα έπρεπε να το σκεφτούμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πω ότι συμφωνώ με τους συναδέλφους και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καβαντά για αυτή την υπέροχη έκθεση. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι μια καλή βάση και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο προανέφεραν και πολλοί συνάδελφοι ότι υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τους στόχους του κανονισμού πρόκειται για διασυνοριακή φορητότητα και όχι για προσβασιμότητα και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι τα περιεχόμενα επιγραμμικών υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν θα πρέπει να έχουν ένα εκούσιο opt in, έτσι όπως προτείνεται εδώ. Και θεωρώ πραγματικά ότι είναι πολύ ικανοποιητικό το γεγονό ότι υπάρχει συνένεση εδώ. Τα σημαντικά σημεία για τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε τι προσεχεί εβδομάδε είναι το θέμα για το πόσο ορίζουμε ε, τι χώρε μέλη διαμονή, καθώ και τα προσωρινά περιεχόμενα, ε, και επίσης πώς θα διενεργούνται οι έλεγχοι. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να τονίσω ότι η Member ε, State of Residence εδώ είναι σημαντικό οι πελάτες να, ε, αναφέρουν την ισχύ μίας διεύθυνσης. Δηλαδή υπάρχει μία διεύθυνση για τον κάθε χρήστη και όχι πολλές διευθύνσεις ή ο συνήθις διαμονή του χρήστη. Έπειτα όσον αφορά την προσωρινή διαμονή, εδώ δεν θα πρέπει να υπάρχει χρονικός περιορισμός, συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε ο κίνδυνος ορισμένες ομάδες στόχο, ε, ορισμένες ομάδες να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, για παράδειγμα οι φοιτητέ Εράσμους, για παράδειγμα. Και όσον αφορά τον έλεγχο του τόπου κατοικίες, θεωρώ ότι είναι σωστή η πρόταση να μην υπάρχουν κλειστοί κατάλογοι ε, κριτηρίων επαλήθευσης και εσείς κύριε Καβαντά το αναφέρατε αυτό γιατί ο κόσμος αλλάζει τόσο ραγδαία που θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία αλλά από την άλλη και μια νομική ασφάλεια βεβαίως. Και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Κέστερ όσον αφορά την τελευταία του παρατήρηση στο θέμα κατά πόσο χρειαζόμαστε μια αυτόνομη αρχή για, την, για τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονισμού. Ε, εδώ έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις και εγώ είμαι επιφυλακτική όπως ο κύριος Κιώστερ γιατί ε, θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί το γραφειοκρατικό άχθο. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν άλλες δυνατότητες για να ελέγξουμε κατά πόσο ε, τηρείται ο κανονισμός ή όχι. Δεν νομίζω θα πρέπει να συσταθεί μια περαιτέρω υπηρεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους ε, ε, εισηγητές των άλλων επιτροπών που συμμετέχουν στη δικασία. Ήδη έχουν αναφέρει πολύ θετικές προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, την νομοθετική διαδικασία σύντομα. Εγώ συμμετείχα ως μέλος της Επιτροπής Εμκο, που νομίζω ότι απάντησε σε πολλά σημαντικά ζητήματα σχετικά με την προσωρινή παρουσία ε, και τα επιπρόσθετα μέσα απαλήθευση. Από τι τροπολογίε ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός ε, σύγκλησης ε, μεταξύ των συναδέλφων για πολλά σημαντικά στοιχεία θεωρώ για τους καταναλωτές, για παράδειγμα η διάταξη φορητότητας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία αύξηση των τιμών, ότι η φορητότητα δεν θα πρέπει να περιορίζεται συμβατικά, για παράδειγμα με ένα χρονικό περιθώριο της φορητότητας. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση και προς αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση στο τοπικό πρόγραμμα, ή τοπικό ρεπερτόριο που θα πρέπει να ε, παρέχεται για τα άτομα με προσωπική παρουσία σε άλλο κράτο μέλο. και συμφωνώ και με τους συναδέλφου που ανέφεραν έναν πιθανό νέο οργανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας. Θεωρώ και εγώ ότι δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Έχω προτείνει μία ρήτρα ε, αναθεώρησης και παρακολούθησης που θα μας επιτρέψει να ε, αναθεωρήσουμε μετά από ένα ευλόγο χρονικό διάστημα και τον κατάλογο των μέσων επαλήθευση, ιδίω ε, και ε, λαμβάνοντα υπόψη και την νομοθεσία για τι μικροψηφίε επιχειρήσει. Με σχόλια τώρα για ζητήματα που θεωρώ ότι εκκρεμούν. Και είναι σημαντικό να τα συζητήσουμε και για την ε, έγκαιρη και ταχεία ολοκλήρωση σε ό,τι αφορά για το νομικό πλάσμα που ε, είναι κάτι το οποίο ανέκυψε και στις άλλες ε, επιτροπές, για τα μέσα επαλήθευσης δεν πρέπει να αναφέρουμε αυτή τη δυνατότητα φορητότητας και να την δυσκολεύουμε, αν θέλετε, περισσότερο από ότι ε, άλλες διαδικασίες που ζητούν επαλήθευση, όπως για παράδειγμα η ψηφοφορία. Δεν ξέρουμε αν χρειάζεται ένα μέσο ή παραπάνω. Εάν το ένα θεωρείται πολύ αδύναμο, τότε θα μπορούσε να λειτουργήσει και ο συνδυασμό δύο μέσων, αλλά και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί αδύναμο. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ έχει βρει μια πολύ καλή λύση. Λέει ότι το ένα μέσο επαλήθευση θα πρέπει να είναι το σύνηθε και μόνο αν υπάρχουν λόγοι αμφισβήτησης αυτού του απλού μηχανισμού, τότε να χρησιμοποιείται ο συνδυασμός δύο μέσων επαλήθευσης. Τώρα, για το tracking, για να ε, καθορίσουμε το ε, κράτος μέλος ε, μόνιμης ε, διαμονής, συμφωνώ με τα όσα είπε ο Κάστα, για, ε, είναι λογικό θεωρώ να μην χρησιμοποιείται το IP για να προσδιορίζεται και η μόνιμη διαμονή και η ε, προσωρινή κατοικία. Και υπάρχουν και στοιχεία προστασίας δεδομένων πρέπει να λεφθούν υπόψη. Ίσως θα ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε μια διεύθυνση IP για να προσδιορίσουμε από πού έχει πρόσβαση αυτό το πρόσωπο στο περιεχόμενο, προσωρινή δηλαδή διαμονή, αλλά μόνο για να του δώσουμε πρόσβαση στο τοπικό ρεπερτόριο, όχι για να ε, προσδιορίσουμε την ακριβή τους ε, θέση ή για να, να αποθηκευθεί μακροχρόνια ε, για την παρακολούθησή του. Δεν θα πρέπει να υπάρξει αποθήκευση των, των διευθύνσεων IP. Τέλος, για το χρονικό θέμα, θεωρώ απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχει ευρεία συνένεση μεταξύ μελών, και όπου και ο κλάδος είχε χρόνο να συνηθίσει την ιδέα αυτού του κανονισμού. Θεωρώ ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα διάστημα έξι μηνών για τη θέση σε ισχύ του κανονισμού και η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν για να συγχρονιστεί με το τέλος των χρεώσεων ε, περιαγωγής, που δεν ξέρουμε τελικά αν θα έρθει, αλλά προς όφελος των καταναλωτών θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ το στεμότερο δυνατόν. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Έχω εντυπωσιαστεί από την ποιότητα της συζήτησης για ένα τόσο τεχνικό θέμα και πολύ καλά το χειρίζονται αυτό το κείμενο οι βουλευτές. Εγώ δεν είμαι καθόλου ειδικό για την ε, για το θέμα της φορητότητας, αλλά θέλω να κάνω κάποιες σκέψεις εδώ. Όταν εξηγούμε τη φορετότητα, ε, ουσιαστικά τι λέμε, ότι υπάρχει ένας συνδρομητής που διαμένει σαν κράτος μέλος και θα μπορεί όταν ταξιδεύει σαν κράτος μέλος να χρησιμοποιήσει τη συνδρομή του. Πολύ συμπαθητικό φαίνεται και μπορεί κάποιο να παρακολουθεί και τις διάφορες ε, σειρές ε, τι τηλεοπτικές. Ε, εγώ δεν με ενθουσιάζει και τόσο, αλλά τέλο πάντων ένας συνδρομητή, ε, θα μπορεί σε άλλο κράτο να παρακολουθεί τη τηλεοπτική σειρά. Έχω τρία σχόλια. Καταρχήν, ο κύριος Καβαδά μας είπε ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να φέρει πρόσθετα κόστος. Όμως μπορούμε να εμποδίσουμε ότι θα υπάρχει προς κόστος. Εγώ δεν είμαι σίγουρος στον επιχειρηματικό κόσμο όταν χορηγούμε μια πρόσθετη υπηρεσία συνήθως ε, την χρεώνουμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να εμποδίσουμε αύξηση του κόστους. Δεύτερη παρατήρηση. Εξηγήσαμε ότι είναι ένα τρόπο να δημιουργήσουμε ένα είδος ε, ενιαίας αγοράς, ψηφιακής αγοράς χωρίς σύνορα. Ξέρετε ότι όλα είναι χωρίς σύνορα προκαλούν τη δυσπιστία μου. Η κατάργηση των σύνορων ε, δεν δίνει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Και πραγματικά εξυπλήσαμε να ακούω ότι η αρχή της εδαφικότητας ε, δεν αμφισβητείται εδώ. Εγώ νομίζω όμως ότι αμφισβητείται και ουσιαστικά την αντικαθιστούμε με μία έννοια πολύ πιο ε, αφηρημένη που είναι το κράτος κατοικίας και εγκαταλείπουμε αυτό που αποτελεί κατά τη γνώμη μου την αρχή της εδαφικότητας, δηλαδή την αρχή της ε, εθνικής προτίμησης. Ε, και αν δεν υπάρχει αυτό, κάθε κράτος θα μπορούσε να χειρίζεται όπως θέλει τις ε, υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου. Όμως εδώ δεν είναι θέμα εγωισμού, αλλά για να υπερασπίσουμε στην περίπτωση της Γαλλίας μια εξαίρεση πολιτιστική που αφορά τη Γαλλία. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Μάλιστα, όταν δίνουμε στη φορητότητα, ε, ουσιαστικά την εικόνα μίας απόλυτης αρχής και λέμε ότι δεν θα περιορίζεται ούτε σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ούτε στα σύνορα. Και μπορούμε εδώ να ευνοήσουμε τελικά τη δημιουργία ολιγοπολίων. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είναι καταστροφική συνέπεια. Και τρίτη παρατήρηση. Είμαι εχθρικός στην επέκτηση της Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία εδώ ότι να δημιουργήσουμε μία νέα ειδική αρχή με ανησυχεί. Όμως δυστυχώς δεν είμαι μόνος σε αυτό το τρίτο θέμα, σε αυτό το τρίτο σημείο που ανησυχώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εκ μέρου τη Σλοβακικής Προεδρίας η κυρία Άγγελα Σομπορτσακοβά. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα και που μας δίνεται και τη δυνατότητα να κάνουμε μία δήλωση εκ μέρους του Συμβουλίου για την πρόταση αυτή. Όπως ε, θα γνωρίζετε το Συμβούλιο ε, έχει, ε, έφτασε σε μία θέση το Μάιο καθώς είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την Ελληνική Προμήθεια, Γενική προσέγγιση είναι τώρα εξισορροπημένο συμβεσμό. Τώρα θέλουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο το συντομότερο. Στο πλαίσιο αυτό η Προεδρία καλωσορίζει την έκθεση τη Γιούρη και σα ευχαριστεί που η ψηφοφορία για την ε, έκθεση αυτή έχει προβλεφθεί για τον Οκτώβριο. Όμω, όπω ακούσαμε σήμερα αναβάλλεται η ψηφοφορία. Αυτό είναι δυστυχέ, καθώς θα καθυστερήσει την θέση ισχύ της πρότασης η Προεδρία. Θα ήθελε λοιπόν να απευθύνει έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει τα δυνατά του προκειμένου να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος το νωρίτερο για να μπορούν να ωφεληθούν οι πολίτες το συντομότερο δυνατόν από αυτή τη σημαντική πρόταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Καβαντά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ γρήγορος γιατί πραγματικά οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις που έκαναν ήταν πολύ χρήσιμες για μένα και πραγματικά συμπληρώνουν αρμονικά το έργο το οποίο ήδη έχει επιτελεστεί. Ε, θα ήθελα ανεκδοτολογικά να πω στον κύριο Μπρατό, όταν πάρετε το αυτοκίνητό και πάτε στο, Βέλγιο, ή στην Ισπανία για 8 μέρες, ε, δεν ε, σταματάτε στα σύνορα. Για αυτό το διάστημα. Είναι το ίδιο ε, ακριβώς συμβαίνει εδώ και εξασφαλίζει πραγματικά και την ε, καλλιτεχνική δημιουργία σε όλες τις ευρωπαϊκές ε, χώρες. Ίσως υπήρξε ένα σφάλμα ερμηνείας, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε. Αλλά είμαι πραγματικά και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, όλους σας ε, και θα πρέπει στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματός μας να συσφίξουμε τη συνεργασία μας ούτε ώστε να συνταχθεί ένα κείμενο το οποίο να είναι ισορροπημένο και το οποίο να συμπεριλαμβάνει κάποιες ε, δικλείδες ασφαλείας κάποιες εγγύσεις. Ωραία λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με το σημείο νούμερο, ε, αριθμό 6 που αφορά τις συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές ε, πτυχές των υιοθεσιών. Και το λόγο έχει κυρία, ο κύριος ε, Ζιέφκα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι πολύ που μπορούμε να προχωρήσουμε τις εργασίες μας σχέση με την έκθεση αυτή και το θέμα αυτής της έκθεσης ε, ε, προσκρούει μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των ε, συναδέλφων και αυτό πάντοτε συμβαίνει με θέματα τα οποία άπτονται των δικαιωμάτων των παιδιών ή αφορούν το οικογενειακό δίκαιο. Και εδώ ισχύει το ίδιο και για αυτή την έκθεση η οποία αφορά τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών και 250 τροπολογίες κατατέθηκαν ε, εδώ και δεν είναι μόνο τροπολογίες από τη δική μας επιτροπή αλλά και από άλλους συναδέλφους. Οι περισσότερες από αυτές τις ε, τροπολογίες συμπληρώνουν το κείμενο ή εισάγουν λύσεις και είμαι ικανοποιημένος γιατί πραγματικά πρόκειται για έναν εμπλουτισμό αυτού του κειμένου και θεωρώ ότι η πλειονότητα των τροπολογιών πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως σας το είπα ήδη, όταν είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσής μου, το πρώτο τμήμα αφορά μια πιο σφαιρική εποπτεία του θέματος των υιοθεσιών. Ε, εδώ παρουσιάζω μια πιο ευρεία, ε, πιο πλατιά εικόνα του ζητήματος της υιοθεσίας. Δεν αφορά τόσο την νομική πτυχή. Αλλά αυτό το τμήμα της έκθεσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί θα πρέπει να περιγράψουμε ε, εξαιρετικά σύνθετα θέματα τα οποία αφορούν τις υιοθεσίε εν γέννη και τις διεθνείς υιοθεσίε ειδικότερα. Αναφέρονται κάποιες ε, ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες θα έπρεπε να ισχύουν όσον αφορά τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών ε, σε σχέση με τη λειτουργία της, με την εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης. Και χαίρομαι που πάρα, οι περισσότερες από τις τροπολογίες που αφορούν αυτό το κομμάτι του κειμένου πηγαίνουν στην κατεύθυνση που ίδιος υιοθέτησα όταν επεξεργάστηκα το σχέδιο έκθεσης. Τα ζητήματα τα οποία συνδέονται με τη διαδικασία της υιοθεσία και με το ουσιαστικό δίκαιο που αφορά το ζήτημα της υιοθεσία δεν μπορούν να ε, ρυθμιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί εναπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των χωρών ε, μελών. Γι' αυτό ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε κάποιους ειδικού κανόνες αυτή τη στιγμή δούμε τις τροπολογίες αυτές και να πάμε προς την κατεύθυνση τροπολογιών επί των οποίων υπάρχει μια γενικευμένη συνένεση, δηλαδή δεν είναι επίμαχες οι τροπολογίες. Και θεωρώ ότι είναι ακριβώς αυτή η προσέγγιση η οποία θα μας επιτρέψει να υιοθετήσουμε ένα κείμενο το οποίο θα μπορέσει μελλοντικά να αποτελέσει τη βάση άλλων εργασιών και είναι ακριβώς αυτό το οποίο αποτελεί τον δικό μας στόχο. Το δεύτερο τμήμα τώρα της έκθεσης ε, υπό τη μορφή παραρτήματος είναι μια πρόταση κανονισμού που θα μπορούσε να ψηφιστεί μελλοντικά και το οποίο θα μπορούσε να προπαρασκευαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση ακριβώς αυτής της έκθεσης ε, επί της οποίας τώρα συζητούμε. Και πιστεύω ότι υπάρχει μια προσδοκία ε, ότι αναμένονται συγγνώμη, κάποιες νομικές τροπολογίες στον ε, τομέα αυτό, δεδομένου ότι οι συμπολίτε μας είναι όλο και πιο κινητικοί και υπάρχουν όλο και περισσότερες διαδικασίες ε, υιοθεσία σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, εκεί όπου είναι εφικτό και ε, στο μέτρο που είναι εφικτό, θα πρέπει πιστεύω να αναζητήσουμε τη δυνατότητα μιας κοινή προσέγγισης και κοινών λύσεων όσον αφορά την ε, αναγνώριση των, ε, εθνικά, ε, ε, των εθνικών υιοθεσιών σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Όσον αφορά την διάρθρωση αυτού του νομικού σχεδίου, έχω βασιστεί σε κανόνες που μας είναι γνωστοί και που λειτουργούν σωστά στους διάφορους τομείς του κοινωτικού δικαίου και με αυτό εννοώ ιδιαίτερος την ε, αμοιβαία αναγνώριση και την ε, εκτέλεση των αποφάσεων ε, υιοθεσιών των δικαστηρίων που υιοθετούνται από, ένα, από μία χώρα και εφαρμόζονται σε μία άλλη χώρα. Ένας μηχανισμός ο οποίος ήδη είναι δοκιμασμένος στην πρακτική και λειτουργεί πολύ καλά. Ε, Βεβαίω έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτή τη στιγμή συζητούμε για μια πρόταση αναγνώρισης των αποφάσεων ε, εγκρίσεων υιοθεσία θα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες που έχουν προβλεφθεί από τις συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όσον αφορά αυτή την πτυχή και προφανώς θα πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι το κείμενο στο οποίο αναφέρεται η αρχή αναγνώρισης των αποφάσεων έγκριση υιοθεσία στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν κυρίως την λειτουργία της κοινή αγοράς. Ενώ σήμερα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πλέον για την ενιαία αγορά εδώ, αλλά αναφερόμαστε σε θέματα τα οποία αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών πρωτίστως και συζητούμε για θέματα τα οποία συνδέονται με, το οικογενικό δίκαιο, το οποίο αναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των χωρών μελών, επαναλαμβάνω. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει εδώ να εφαρμοστεί η αρχή ε, ε, της ε, λογικής και να δημιουργηθεί μια πρόταση η οποία ε, θα κάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να την υιοθετήσει για να προτείνει ένα νέο νομικό κείμενο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επαγρυπνήσουμε ώστε στη δική μας έκθεση να συμπελθούν κάποιες πτυχές οι οποίες ε, δεν θα έχουν σαν αποτέλεσμα απλούστατα να απορριφθεί η πρόταση αυτή και το θέμα αυτό να φύγει από το τραπέζι για πολλά χρόνια στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ήταν απευκταίο. Και θα ήθελα να πω το εξή. Για ποια νομικά εργαλεία μιλούμε εδώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λογικά κάποια δοκιμασμένα εργαλεία. Βεβαίως υπάρχουν, ε, δυστυχώς υπάρχουν ε, Πολλέ τροπολογίε ή μια ομάδα τροπολογιών που δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Η πρώτη τέτοια ομάδα τροπολογιών αφορά τη θέση εν αμφιβόλο της ρήτρα της δημόσιας τάξης. Η ρήτρα αυτή της δημόσιας τάξης ε, παρουσιάζεται σαν ένα μέσο ε, εφαρμογής διακρίσεων. Και νομίζω ότι αυτό είναι εντελώς παράλογο. Κυρίες και κύριοι, η ρήτρα αυτή είναι μια βασική αρχή του διεθνούς, ε, του ιδιωτικού δικαίου. Αυτή η ρήτρα υπάρχει και στον ε, κανονισμό των ε, Βρυξελών και σε, άλλες, και σε άλλους κανονισμούς που αφορούν πολλά θέματα κληρονομιάς ε, και η ρήτρα αυτή υπάρχει και σε διεθνείς συμβάσεις ιδιαίτερο στην ε, σύμβαση την οποία αναφέρομαι στη δική μου έκθεση, δηλαδή τη σύμβαση του 1000, της Χάγης του 1993 που αφορά την προστασία των παιδιών και την συνεργασία στο θέμα των διασυνοριακών ε, υιοθεσιών. Πώς λοιπόν μπορούμε να αφισβητήσουμε αυτήν ακριβώς τη ρήτρα. Το ίδιο ισχύει και για ένα άλλο στοιχείο, το οποίο επίσης ε, αναφέρει σε ορισμένε τροπολογίε που έχουν κατατεθεί, δηλαδή την άρνηση αναγνώρισης των αποφάσεων ε, υιοθεσία, έγκρισης υιοθεσία ή τη δυνατότητα να προσφύγει κανείς αυτή τη στιγμή υπάρχει απόρριψη της δυνατότητας αναγνώρισης. Εάν δεν υπάρχουν, υπάρχει δυνατότητα προσφυγή σε ένδικα μέσα, δεν είναι δυνατόν να ισχύσει ο κανονισμός και απλούστατα το κείμενο αυτό μπορούμε να το πετάξουμε στον κάλαθο αχρήστων και να το ξεχάσουμε χωρίς να αναφέρουμε το γεγονός ότι μια τέτοιου είδους ε, προσέγγιση ε, απλούστατα, είναι, αντιβαίνει στην αρχή της ε, καθολικής ε, πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Είναι, αντιβαίνει στην ε, αρχή του δικαιώματος προσφυγής ένδικα μέσα που πάντοτε προβλέπεται σε, εντός μιας νομικής διαδικασίας και που είναι ισόφαλος όλων των ενεχόμενων μερών προφανώς θα πρέπει να ε, δούμε την ε, φύση εδώ του θέματος. Γι' αυτό είναι ακριβώς δύσκολο να διακρίνουμε τα ιδεολογικά από τα νομικά θέματα, αλλά παρόλα αυτά κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να πάμε πέρα από τα όρια μιας ιδεολογικής προσέγγισης στο κείμενο αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε λύσεις που θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές ε, για όλους. Ήδη έχουμε εργαστεί πολλών θεμάτων στους κόλπους της Επιτροπής και συχνά είπαμε ότι θα αξίζει περισσότερο να κάνουμε ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση παρά να κάνουμε ένα μεγάλο διακελισμό, διασκελισμό πολύ μακριά. Ούτε σωστή, αλλά μην μπορούν να μας ακολουθήσουν. Γι' αυτό προσωπικά είμαι κατά τροπολογιών που κατατέθηκαν και που αφορούν το θέμα της ε, ε, κοίησης, της παρένθετης κοίησης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα, το οποίο θα χρειαζόταν ένα άλλο κείμενο. Ε, χρήση μεγαλύτερης προσοχής και δεν ήταν το να συμπεριληφθεί έτσι σε μια τέτοια έκθεση. Γι' αυτό είναι κατά όλων αυτών ε, τροπολογιών που αφορούν τις παρένθετες μητέρες. Επίσης θα ήθελα να παρουσιάσω τις συμβαστικές τροπολογίες, τις δικές μου. Πολλές τροπολογίες έχουν κατατεθεί, γι' αυτό θα ήταν καλό την ε, προσεχή εβδομάδα να έχουμε μία ε, συνάντηση εργασίας όπου θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στις εργασίες μας χωρίς να αναφέρουμε στο σύνολο των ετοιμάτων της Επιτροπής. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια τέτοια εργασία και ελπίζω να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το κείμενο αυτό, να θέσουμε στις ψηφορίες στην προσεχή συνεδρία του Νοεμβρίου, ούτω ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της, ε, ε, του έτους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες και συνέβαλαν στις εργασίες ε, αυτές. Ε, Παρουσιάζω και στις παρατηρήσεις. Είμαι ανοιχτός προς τα σχόλια όλων των συναδέλφων και είμαι ευτυχής και για τη συνέχιση της εργασίας, τελευταία φάση εργασιών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσφεύκα για την παρουσίασή του και για την προσέγγιση που ακολούθησε. Για την προθυμία του να συζητήσει αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Αν δούμε τον υψηλό αριθμό τροπολογιών, καταλαβαίνει κανείς ε, πόσο λεπτό είναι αυτό το ζήτημα. Όταν εγώ ήμουν νομικός, ασχολήθηκα επισταμένως με τις διεθνεί υιοθεσίε, ξέρω ποιε είναι οι δυσκολίε και είναι πολύ σημαντικό μέσω της νομοθεσίας που προσπαθούμε να καταρτήσουμε να έχουμε τελικά κάποιες ε, κατευθυντήρες γραμμές για μελλοντικές τροποποιήσει τροποποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα, βασικό μας μέλημα θα πρέπει να είναι το συμφέρον του παιδιού. Ακόμα και αν θεσπίσουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τις τρίτες χώρες που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο συγκεκριμένα Ελβετία και Νορβηγία, και την αναγκαιότητα να εισάγουμε σε αυτή την εξίσωση αυτές τις πτυχές που συνδέονται με τα, με τα δικαιώματα του παιδιού. Δεν θέλω να αναφερθώ στο ιστορικό. Ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα με τις διεθνεί υιοθεσίε γιατί δεν ακολουθούν τους κανόνες που προσπαθούμε να επιβάλλουμε εδώ. Δεν νομίζουμε ότι ένα παιδί είναι ιδιοκτησία του κράτους. Ε, ανήκει στους γονεί του. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Από την άλλη, με προβληματίζει ιδιαίτερα το τι συμβαίνει μετά την υιοθεσία σε ένα κράτος μέλος. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν μετά την υιοθεσία ή εάν οι γονεί στο κράτος μέλος δεν έχουν πλέον γονεϊκά δικαιώματα και το παιδί δοθεί προς υιοθεσία εντός του κράτους μέλους και πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι σε μία υπόθεση στην Μεγάλη Βρετανία, όπου είχαμε Ρουμάνους γονείς που έμεναν στην ε, Μεγάλη Βρετανία, έχασαν τα γονεϊκά τους, δικαιώματα, χωρίς να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα. Τα παιδιά τους λοιπόν δόθηκαν προς υιοθεσία σε ένα ομόφυλο ζευγάρι. Στη Ρουμανία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν ε, αναγνωρίζεται ο γάμος μεταξύ ομοφύλων. Επομένω, προφανώ δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοια υιοθεσία στη Ρουμανία και νομίζω ότι δεν πρέπει να το γνωρούμε αυτό. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε το παιδί που δίνεται για υιοθεσία να αναπτύσσεται μέσα στο ίδιο πολιτιστικό ε, και θρησκευτικό πλαίσιο όπως στη χώρα από την οποία προέρχεται. Ιδάλλως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τήρηση του, των συμφερόντων του παιδιού. Νομίζω τελικά ότι θα καταλήξουμε όμως σε μια ισορροπημένη λύση, γιατί βέβαια τα κράτη-μέλη ε, εδώ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα. Όμως κάποια ζητήματα θα πρέπει να τα καθορίσουμε και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, γι' αυτό τα συζητάμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια έκφραση αλληλεγγύης. Ευχαριστώ, κυρία Χαπταλά. Ευχαριστώ πολύ. Ορισμένες ερωτήσεις για τις προτάσεις ε, ως προς το άρθρο 6 για την άρνηση αναγνώρισης. Να σας το διαβάσω. Η αναγνώριση αθεσίας, απόφασης μάλλον προς αθεσία, μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν αυτή η αναγνώριση ε, προδήλως αντιβαίνει στις αρχές δημοσίας τάξης του κράτους μέλους. Η δημόσια τάξη είναι η πλέον ευρεία και αφηρημένη έννοια που χρησιμοποιείται στην νομοθεσία. Θα ήταν καλό να κατανοήσουμε σε τι είδους καταστάσεις αναφερόμαστε εδώ. Αλλιώς μπαίνουμε λίγο σε μια θεά ζώνη, αν βάλουμε τέτοιου είδους όρους στην νομοθεσία μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γοζιέ, κάτι τεχνικό θέλετε να θέσετε. Συνήθω δίνουμε τον λόγο στου κοιόδη τη κι οπότε περίμενα να το πάρω, αλλά τέλο πάντων σα ζήτησα το λόγο ω κοιόδη εισηγήτρια για του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ε, παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρο. Λοιπόν, ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Είναι όντω σημαντικό ο σκοπό αυτό, να επιτρέψουμε την αυτόματη αναγνώριση των διεθνών υιοθεσιών αρκετά συχνά βλέπουμε προβληματικέ ε, καταστάσει και υποθέσει σε τέτοιου είδου διασυνοριακέ υιοθεσίε, είτε μέσω των μέσων ενημέρωση, είτε και στο Κοινοβούλιο. Επομένω, είναι σημαντικό να λύσουμε αυτό το ζήτημα και γι' αυτό απαιτείται Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και πάλι, λοιπόν, ευχαριστώ τον εισηγητή. Στόχο, είναι η διασφάλιση της ε, ασφάλεια δικαίου, αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και των γονέων. Στηρίζω λοιπόν την έκθεση, ιδίω σε ό,τι αφορά αυτόν τον στόχο ε, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα κυρίαρχα δικαιώματα του παιδιού. Ε, στο επίκεντρο να τεθεί αυτή η αρχή λοιπόν στις αποφάσεις υιοθεσιών και τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν τα δικαιώματα του παιδιού ε, ως προς την ελεύθερη έκφραση και να λαμβάνεται υπόψη γνώμη του τελικά. Βεβαίως ε, αυτό το κείμενο ε, προκαλεί το ενδιαφέρον, πολλές τροπολογίες και εγώ εξέφρασα με δυσαρέσκεια κάποιες ε, προτάσεις που θεωρώ ότι θα πρέπει να απορρίψουμε. Ιδίω όλες τις τροπολογίες που θέλουν να αφαιρέσουν κάθε νόημα και κάθε περιεχόμενο από το κείμενο, το οποίο εμεί χρειαζόμαστε κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχουν χώρο στο κείμενο. Καλό θα είναι να μην μπούμε σε άλλα ζητήματα που δεν μας αφορούν εδώ. Πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς στο ζήτημα το οποίο είναι η διασφάλιση του κυρίαρχου ε, συμφέροντος του παιδιού. Και όπως αναφέρει και ο εισηγητής, τροπολογίες που θέλουν να υποτάξουν το κυρίαρχο δικαίωμα του παιδιού στην ε, ε, εθνική δημόσια τάξη. Για μας δεν είναι αποδεκτό αυτό. Πρέπει το συμφέρον του παιδιού να τεθεί στο επίκεντρο τη συζήτηση. Έχω υποβάλει πολλές τροπολογίες, κάποιες ε, που ε, εξαλείφουν οποιαδήποτε δυνατότητα διακρίσεων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό ε, για το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να διασφαλίζεται στο κείμενο. Κλείνοντα, ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή και σίγουρα θα έχουμε πολύ υποκατηματικέ ανταλλαγέ απόψεων κατά την προετοιμασία του τελικού κειμένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τζεύσκα για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις ε, για όλες αυτές τις τροπολογίες που ξεπερνούν τις 200. Πιστεύω ότι ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές ε, θα έχουν κατά νου το στο συμφέρον του παιδιού και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να δεχτείτε τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν ε, με την υθεσία του παιδιού στα πλαίσια της βιολογικής οικογένειας. Έχουμε, έχω στείλει πολλές τροπολογίες για την κατάρτιση και τη συνεργασία μεταξύ δικαστών, ε, νομικών, κυβερνητικών υπαλλήλων και κοινωνικών λειτουργών που θα συμμετέχουν σε αυτές τις διασυνοριακές διαδικασίες. Επίσης, οι κυβερνητικοί φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν και να ξεπεράσουν μία σειρά διαφορών. Και εγώ θα ήθελα το πιστοποιητικό υιοθεσία να είναι σε πολλές γλώσσες έτσι ώστε να μην έχουμε και κόστος για την μετάφραση. Ο κ. Λεμπρετών, ευχαριστώ πρόεδρε η σύμβαση της ε, Χάγης ε, του 1993 είναι μια πολύ καλή σύμβαση και ουσιαστικά έχει πλεονεκτήματα, αφενός οργανώνει μια διεθνή συνεργασία και αφετέρου σέβεται και την κυριαρχία του κάθε κράτους. Η πτυχή της συνεργασίας έχει να κάνει με την αναγνώριση από κάθε κράτος των ηθεσιών που γίνονται στην επικράτεια άλλων κρατών που υπογράφουν και ο σεβασμός ε, της ε, εθνικής κυριαρχίας ε, γίνεται διατηρώντας ουσιαστικά την δημόσια τάξη, γιατί ουσιαστικά πρέπει να γίνεται σεβαστή η δημόσια τάξη. θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ό,τι αφορά την αναγνώριση των Παρ' ε, Παρόλα αυτά, δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν καλές προθέσεις, όμως ε, φοβάμαι μήπως έχουμε αρνητικές συνέπειες και θα αναφέρω δύο. Καταρχήν, ότι τελικά θα αμφισβητήσουμε την τήρηση της δημόσιας τάξης. Αυτό έχει γίνει ήδη σήμερα προφορικά και κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ περισσοδεδεμένο σε αυτό. Εδώ μιλάμε για το θέμα της εθνικής κυριαρχίας για μια ακόμα φορά. Προσπαθούμε να έχουμε ενοποίηση και ομοιομορφία ενό τομέα, ενώ τα κράτη-μέλη θέλουν να διατηρήσουν περιθώριο ελιγμών και επίσης ε, μέσω των τροπολογιών θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μέσα και το θέμα της ε, κοίησης ε, για κάποιο άλλο άτομο και αυτό είναι εντελώ διαφορετικό και πραγματικά με ξέπληκε που σας άκουσα σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε την έκφραση το ανώτατο συμφέρον του παιδιού, το βαλτιστό συμφέρον του παιδιού. Δεν είμαι εχθρικό απέναντι στην εκφρασία αυτή, Όμω, προσοχή. Είναι τελείω εντουβεντελιστική αυτή η φράση. Εγώ ε, παρατηρώ ότι η σύμβαση τη Χάγη δεν έχει γίνει μόνο προ το συμφέρον του παιδιού, αλλά και προ το συμφέρον των οικογενειών και τη οικογένεια. Να μην ξεχνάμε την τύχη αυτή. Κυρία Χαουτάλα, να ευχαριστώ. Ήδη κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, άκουσα το, δύο φορέ για το θέμα των παρένθετων μητέρων και θα ήθελα να πω ότι είναι εντελώ ξεχωριστό θέμα, αλλά παρόλα αυτά έχει να κάνει με το διεθνέ ιδιωτικό δίκαιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αρχίσει να το διερευνά αυτή η Επιτροπή και όταν επισκεφθήκαμε πέρσι το χειμώνα μία συνάντηση για τη Σύμβαση της Χάγης ε, και για το Διεθνές Δίκαιο. Ακούσαμε και πίσω εμπειρογνώμενες, οι μας ε, ε, είπαν ότι γνωρίζουν ότι είναι σημαντική η δουλειά τους για τη δουλειά της δικής μας Επιτροπής. Επίσης, επειδή υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, όπως η παράγραφος που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο μιας μακροσκελής έκθεσης για τετήσει ανθρώπινα δικαιώματα πριν μισό έτος, νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να διερευνήσουμε αυτό το θέμα πολύ σοβαρά γιατί θα πρέπει να ρυθμιστεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η... το θέμα της παρένθετης ε, μητέρας. Ε, νομίζω εδώ πάντοτε θα πρέπει να, της παρένθετης κοίησης, θα πρέπει να έχουμε στο προσκήνιο το συμφέρον του παιδιού. Γιατί ε, πράγματα τα οποία είναι δύσκολα και ευαίσθητα παρόλα αυτά λαμβάνουν χώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να ρυθμιστούν μέσω του αστικού δικαίου στην Ευρώπη. Ωστόσο, εγώ ήθελα να πάρω το λόγο ε, είναι διαφορετικός. Θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Ε, Την τελευταία πράσινη εβδομάδα υπήρξε η Eurolat και υπήρξαν και ορισμένοι βουλευτές ε, αυτής της επιτροπής που πήγαν στο Μοντεβίδεο και εκεί ασχολήθηκαν με το εξής θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις υιοθεσίες και είναι προφανές στην Λατινική Αμερική υπάρχουν πολλές απαγωγές παιδιών. Είναι μη ξεκάθαρη προέλευση των παιδιών τα οποία στη συνέχεια υιοθετούνται. Και ήταν ένα εντελώ πιστικό εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίο είπε ότι μέσω των τεστ DNA είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αυτό με μεγάλη ακρίβεια. Θα πρέπει λοιπόν οι δοκιμές τα τεστ αυτά, το DNA, να συμπεριληφθούν ε, στο διεθνές ε, δίκαιο. Ε, υπάρχουν ε, πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ήταν εκεί και οι οποίοι θεώρησαν ότι ήταν μια πολύ λογική σύσταση και ίσως θα έπρεπε να συσταθεί μια έκθεση πρωτοβουλίας. Δεν ξέρω αν είναι δεδειγμένη εδώ η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Και μια και έχουμε όμω σήμερα στην ημερήσια διάταξη θέματων των υιοθεσιών και ο κ. έκανε μια καλή έκθεση ε, θα ήθελα να θέσω το ερώτημά μου κατά πόσο είναι δυνατόν στο στάδιο αυτό να προετοιμάσουμε μια σχετική τροπολογία για την Ολομέλεια ή τελικά ε, ποια θα είναι η διαδικασία μέσα στις οποίες θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα που σας ανέφερα και το οποίο πολιτικά πραγματικά είναι αδιαμφισβήτητο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπελσερό. Ναι, ε, συμφωνώ απολύτως ε, με το όσα είπε η κυρία Ρέγκνερ. Ε, ήδη έχουμε ανταλλάξει, ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις εκεί και έστω και αν το, θέμα αυτών των τεστ, και αυτά τα τεστ, αυτά καθ' αυτά είναι σοκαριστικά, παρόλα αυτά θα πρέπει να γίνουν. Εγώ υιοθέτησα ένα παιδί από τη Ρουμανία και όταν μου παρουσίασαν το παιδί ε, ε, ρώτησα κατά πόσο συμφωνούσε η μητέρα του. Ε, πρόκειται για ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Βέβαια, η έκθεση του κ. Ζήφσκα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Μπρετόν. Εγώ αν ήμουν ευρωσκεπτικίστρια στη, ε, στη ζωή μου θα έλεγα ότι ε, τα ανθρώπινα όντα θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πρόκειται για το θέμα ακριβώ αυτής της έκθεσης. Και εδώ είναι απολύτως ενδεδειγμένο το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στη Γαλλία υπάρχει, υπάρχουν δύο μορφές υιοθεσίας. Η απλή, όπου οι γονείς ε, δεν έχουν όλα τα δικαιώματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάση περιπτώσει για την έκθεσή σας. Ε, euh, Πολύ γρήγορα, Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Ζιευκά για το βάθος το προβληματισμό του και την ευαισθησία που προκύπτουν. Θα ήθελα να στηρίξω όσα είπε η κυρία Ρέγκνεν και η κυρία Περσερόν. Έχουμε πολύ σημαντικές σχέσεις με χώρες όπως η Ρωσία και στο εσωτερικό των κρατών μελών είχαμε μεγάλη κινητικότητα παιδιών. Κάποιος μίλησε για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Όμως ε, είμαστε κάπως αδιάφοροι. Θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το εξή δράμα. Του χάρη αυτά που έγιναν πριν 25-30 χρόνια στη Λατινική Αμερική αναφέρθηκε το Μοντεβιδέο αλλά εγώ το είδα αυτό το θέμα και στην Αργεντινή, στη Χιλή, στη Βραζιλία, στην Κολομβία. Πρόκειται λοιπόν για ένα παγκόσμιο πρόβλημα που πουθενά δεν έχει λυθεί και υπάρχει απόλυτη σιωπή. Πρόκειται για δεκτορίες που είτε εκτόπισαν, μετατόπισαν τα παιδιά, είτε σκότωσαν τους γονείς ή ολόκληρες οικογένειες ή υιοθέτησαν με τη βία άλλα παιδιά. Και δεν βρίσκω άλλη λύση παρά την εξέταση DNA για να δούμε ουσιαστικά ε, αν φυσικά το παιδί το επιθυμεί να μπορεί να έχει δικαιώματα νόμιμα απέναντι στην βιολογική του οικογένεια. Και εδώ θα ήθελα να ξαναναφέρω την ιδέα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τα παιδιά. Ουσιαστικά είναι ένας ε, από τους ε, τομείς που είναι τόσο εθνικοποιημένοι και δημιουργούνται και αδικίες. you very uh, I felt from Ευχαριστώ. Κάποιες ε, από τις παρατηρήσεις του κυρίου Λεμπρετών κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Γιατί όπως γνωρίζετε η συζήτηση θα μπορούσε να δώσει μια ψευδή εντύπωση ότι η εθνική κυριαρχία ουσιαστικά <laughs> προσαρτάται μόνο σε ένα κράτος. Και το σημερινό δόγμα για το κράτος και το δίκαιο, όπως έχει επιβεβαιωθεί και από πολλά συνταγματικά δικαστήρια, υπάρχουν πολλά επίπεδα, περισσότερα επίπεδα ε, εθνικής κυριαρχίας, παραδείγματος χάρη υπάρχει κυριαρχία του λαού, κυριαρχία, μπορεί να αποφασίσει παραδείγματος χάρη ο λαός και μπορεί να υπάρχει λοιπόν μετακύληση της έννοιας της κυριαρχίας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να το εξετάσουμε. Δεν ε, αφορά μόνο το επίπεδο του κράτους. Τώρα, για την Κομισιόν κυρία Ντελούκα. Ε, Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την πλήρη έκθεσή του για αυτό το ευαίσθητο θέμα. Από τα κράτη-μέλη έχουν αποκλίνουσες απόψεις. Επομένως, η Κομισιόν πιστεύει ότι είναι σημαντικό για ποια θέματα μιλάμε, δηλαδή την διασυνορική αναγνώριση εντολών υιοθέτηση ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωση και συγκεκριμένα να συμφωνήσουμε για το τι είναι εκτός του πεδίου εφαρμογή. Γιατί η διασυνορική αναγνώριση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ένα θέμα υιοθεσία χωρίς ε, ε, τη συνένεση, η καταναγκαστική υιοθεσία που γίνεται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με τρίτες χώρες όπως η Νορβηγία. Ε, δεν είναι και περί παρέμφετων μητερών, ούτε περί εμπορίας παιδιών, ούτε περί ουσιαστικού εθνικού δικαίου για την υιοθεσία, το οποίο μπήπτει στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους ούτε μιλάμε για διασυνοριακές υιοθεσίε, γιατί η διασυνοριακή υιοθεσία είναι μια υιοθεσία όπου οι γονείς ε, και το παιδί είναι σε διαφορετικά κράτη. Εδώ μιλάμε για την εξή περίπτωση. Μια εθνική υιοθεσία λαμβάνει η χώρα σε ένα κράτος μέλος και κατόπιν οι θετοί γονείς θέλουν να αναγνωριστεί αυτή η υιοθεσία από ένα άλλο κράτος μέλος και μιλάμε για το πρόβλημα που δημιουργεί η έλλειψη αυτή τη αναγνώριση για του γονεί. Παραδείγματο χάρη για την ελευθερία μετακίνηση του εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για το παιδί, γιατί το νομικό του καθεστώ δεν έχει αναγνωριστεί. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν της συζήτησης. Τα υπόλοιπα θέματα φανώς είναι πολύ σημαντικά αλλά η Κομισιόν ε, δεν θεωρεί ότι πρέπει όλα να τα βάλουμε σε μία έκθεση. Γιατί όπως ε, είπαν και άλλες επιτροπές, ε, δηλαδή το θέμα της υιοθέτηση χωρίς συνένεση κτλ. Πρέπει να προσδιορίσουμε και ποιο είναι το θέμα. Κομισιόν εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά την πρόταση του εισηγητή. Ευχαριστώ. Thank you as well. Uh, Mr. Ευχαριστώ κύριε Ζβεύκα. Έχει τελευταίο στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Σας ευχαριστώ για τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχόλιά σας. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τελοκόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί σε μερικές προτάσεις συνοψίσατε ε, όλα όσα βρισκόνται στο επίκεντρο αυτής της έκθεσης. Αυτό ακριβώ που είπατε μόλις τώρα είναι η σύνοψη της ε, ουσίας ε, της έκθεσης και αυτό θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε και τις εργασίες μας. Και σας ευχαριστώ. Όλα τα σχόλια μας ήταν ενδιαφέροντα. Ο κύριος Λεμπογατού, σέβομαι την άποψή σα παρότι διαφωνώ κάθετα μαζί σας. Δεν θέλω λοιπόν να αντιδράσω και να σχολιάσω περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά την ε, δημόσια τάξη, η κυρία Χάουταλα αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα. Ε, να σας υπενθυμίσω μόνο ότι έχει εκπονηθεί μελέτη σε αυτό το ζήτημα από έναν καθηγητή ε, που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά τέλο πάντων είναι καθηγητή τη Σορβόνη και μπορείτε να την βρείτε στη γραμματεία αν θέλετε αυτή τη μελέτη. Και να σα υπενθυμίσω και πάλι ότι πρόκειται για μια βασική έννοια στο διεθνέ δίκαιο. Είναι μια αρχή την οποία βρίσκουμε ε, στα κείμενα που έχουμε υιοθετήσει ε, αλλά και στα κείμενα που τώρα εξετάζουμε. Επενθυμίζω αυτό που σας ζήτησα στην αρχή της παρέμβασής μου. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε συγκρατημένοι ως προς τη συμπερίληψη όλων των σημαντικών στοιχείων μέσα στην έκθεση. Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικά τα όσα αναφέρατε. Πρόκειται για θεμελιώδει ε, αρχέ ε, ω προ τα δικαιώματα του παιδιού, ε, σε ό,τι αφορά τις ε, αναγκαστικές υιοθεσίε ή τις ε, παράνομες υιοθεσίε, τις παρένθετες μητέρες, διεθνή συνεργασία, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά που είπατε και μπορούμε να τα συζητήσουμε, όμως ας προσπαθήσουμε να περιοριστούμε στον δικό μας τομέα αρμοδιοτήτων. Ποιες είναι οι δικές μας αρμοδιότητες, τι θέλουμε ακριβώς να ρυθμίσουμε εμείς για να βελτιώσουμε τα πράγματα, να έχουμε μια καλύτερη λύση σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η μοναδική μου πρόθεση. Τα υπόλοιπα μπορούμε βεβαίως να τα συζητήσουμε εκ νέου. Ε, και το ζήτημα που ανέφερε ο κύριος ε, Πρόεδρος, ε, με το οποίο συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την προσέγγιση που αναφέρατε, ε, την κυριαρχία, τη δικαιοδοσία, ε, τα διάφορα επίπεδα, διάφορες διαστάσεις. Γιατί κάποιες φορές ε, εξετάζουμε με πολύ περιορισμένο τρόπο αυτό το ζήτημα. Υπερθυμίζω και πάλι την πρόταση να διοργανώσουμε μία συνάντηση εργασίας την επόμενη εβδομάδα. Λαμβάνοντα όχι μία μινιμαλιστική, μάλλον πιο ρεαλιστική προσέγγιση και έτσι θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Έτσι βέβαια δεν κλείνουμε την πόρτα σε, μία, ε, σε βάθος συζήτηση στη συνέχεια, αλλά για να προστατεύσουμε, να σώσουμε αυτή την πρόταση, για να έχει δυνατότητες και πιθανότητες υλοποίησης ως ε, νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας είμαστε λοιπόν πιο συγκρατημένοι και να μην ε, συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα στοιχεία στην πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσαμε το σημείο 6. Πάμε στο σημείο 7. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. Το λόγο έχει ο κύριος Καβαντά. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την ε, οδηγία σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων του 1996 έχει ως ε, σκοπό να εισαγάγει ορισμένα νέα μέτρα να ε, εξαλείψει ορισμένες αθέμητες πρακτικές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οποίες καταγγέλουν αρκετά με συστηματικό και έντονο τρόπο. Θα ήθελα εδώ να επενθυμίσω τις τρεις ε, βασικές τροποποιήσεις που θέλουμε να σαγάγουμε εδώ. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την άμεση απόσπαση ε, εισάγεται η αρχή της ε, αποζημίωσης ε, που αντικαθιστά τον κατώτατο μισθό. Πλέον έχουμε την αποζημίωση ή αμοιβή που θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους που θα υπάρχουν στον ίδιο τόπο και διεξάγουν τις ίδιες εργασίες. Βάσει λοιπόν του τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται, κρίνονται. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν την ίδια αμοιβή για τους εργαζόμενους ε, και στις ε, αλυσίδες υπεργολαβίας. Το δεύτερο σημείο, ε, η πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί τους κανόνες για την εποχική εργασία. Η Συνθήκε ε, που θα επιβάλλονται στις διασυνοριακές επιχειρήσεις για την προσωρινή απασχόληση, όπου δηλαδή ε, αποσπώνται εργαζόμενοι ε, σε άλλη χώρα, θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με τους εργαζόμενους στο εθνικό πλαίσιο απασχόλησης και έτσι να υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων. Το τρίτο, πρόταση περιορισμού της διάρκειας της απόσπασης του εργαζομένου στους 24 μήνες. Εάν υπερβούμε αυτό το χρονικό περιθώριο, το κράτος μέλος εργασίας θα θεωρείται μόνιμος τόπος εργασίας του εργαζομένου. Υπάρχει λοιπόν ο χρονικός περιορισμός. Όπως ξέρετε, το κείμενο αυτό αποτέλεσε αντικείμενο ε, Μια διαδικασία κίτρινη κάρτας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει ε, την πρότασή τη. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ήταν ότι τα ε, επιχειρήματα που κατέθεσε η άλλη πλευρά δεν ευσταθούσαν και εγώ να προσθέσω ότι μάλλον συμφωνώ με αυτό το συλλογισμό. Η αναθεώρηση θεωρήθηκε απαραίτητη από όλους ε, αλλά και, και για τις μεγάλες επιχειρήσεις και από τις μικρές επιχειρήσεις και ε, οι ψηφοφόροι είδαν ότι υπάρχει ένα σημαντικό σημείο ανισότητας σε ό,τι φορά τη μετατόπιση ε, εργαζομένων εθνικών επιχειρήσεων και πολύ σημαντική αδικία. Ήρθε λοιπόν πλέον η ώρα να τροποποιήσουμε αυτό το κείμενο του 1996. Είναι λοιπόν απαραίτητη η αναθεώρηση, επίγουσα, εξαιτία των καταχρήσεων που έχουμε παρατηρήσει και έχουν πολύ δυσμενείς συνέπειες και για τις ε, επιχειρήσεις ε, ταχυδρομικής θηρίδας και μόνο, που είναι δηλαδή μια απάτη ουσιαστικά, που ηθικά είναι παράνομη, νομικά προς το παρόν γίνεται αποδεκτή. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε. Και το πλαίσιο που διέπει την μετατόπιση των εργαζομένων ε, έχριζε βελτίωση και θεωρώ ότι πρέπει να ε, θεσπιστεί τώρα με καλύτερο τρόπο. Βεβαίω θα πρέπει να περιορίζονται οι ελευθερίες ε, που προβλέπονται από τις ε, συνθήκες. Ε, πιο συγκεκριμένα την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την ελευθερία εγκαθίδρυσης και εγκατάστασης και την παροχή υπηρεσιών. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε αυτή την πολύ χρήσιμη μετακίνηση, απλώς θέλουμε να διαμορφώσουμε μια βάση ισότητας και να αποφύγουμε τις τρευλώσει που είναι καταστροφικές και για την οικονομία και για την απασχόληση και για τις επιχειρήσεις σε ένα βαθμό. Τέλος, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ε, μπούμε στα χωράφια της Επιτροπής Απασχόλησης. Η δική μας Επιτροπή είναι αρμόδια για την ερμηνεία και την εφαρμογή ε, του ευρωπαϊκού δικαίου. Γι' αυτό θα ήθελα στη γνωμοδότησή μου να συμπεριλάβουμε και ορισμένα σχόλια σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση της ε, πρότασης και διασύνδεσή της με τον κανονισμό Ρώμη 1 και τη συμβατότητά του, τη συμβατότητα μεταξύ των δύο κειμένων μάλλον. Το προσωρινό χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Σήμερα το πρωί όλο για χρονοδιαγράμματα σας λέω. Ε, 28 ε, Νοεμβρίου παρουσίαση του προσχεδίου, μέχρι 7 ε, Δεκεμβρίου υποβολή τροπολογιών και υιοθέτηση στην ε, Επιτροπή μας τον Φεβρουάριο του 2017. Προς ενημέρωσή σας, η, απασχόληση, η Επιτροπή Απασχόλησης έχει αποφασίσει να ψηφίσει τον Απρίλιο του 2017 Επομένω, νομίζω ότι βγαίνει ωραία το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ και είμαι και πάλι στη διάθεσή σας ε, να εργαστούμε αρμονικά ε, με όλους όσοι θέλουν να βελτιώσουμε την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λοτόφσκι έχει το λόγο. E, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω μερικά λόγια για το θέμα αυτό με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Πιστεύω ότι η αλλαγή της ε, οδηγίας που προτείνεται από την Επιτροπή μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες νομικές ε, αμφιβολίες ε, και χωρίς ένα νομικό έλεγχο δεν θα γνωρίζουμε κατά πόσο οι αλλαγές δεν θα έχουν επιπτώσει στη διαφάνεια του ευρωπαϊκού δικαίου. Υπάρχουν κάποια προφανή ελλείμματα ε, γιατί διαφωνεί με τους θεμελιώδεις κανόνες της συνθήκης, ιδιαίτερα στην αρχή της επικουρικότητας. Και 11 χώρες ε, κίνησαν τη δικασία με κίτρινη κάρτα. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες ενστάσεις. Αυτή η αρχή είναι πολύ σημαντική προκειμένου να φτάσουμε σε μια ισορροπία μεταξύ θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών κυβερνήσεων το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ε, το ζήτησε τον ε, σεβασμό αυτής της ε, αρχής. Επίσης, η Επιτροπή δεν τήρησε ορισμένες υποχρεώσεις που είχε δεσμευθεί να αναλάβει. δεν υπήρξε κοινωνική διαβούλευση και δεν έγινε οικονομική μελέτη όσον αφορά τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών. Τα αποτελέσματα της ε, τροποποίησης της οδηγίας ε, δεν είναι παρά ε, ευσεβείς πόθη για ορισμένες χώρες. πολλές ε, επιχειρήσεις απλούστατα, ε, εάν ισχύσει αυτό, θα πάψουν να υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να το αγνοήσουμε. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε το νομικό χάος που θα μπορούσε η τροποποίηση αυτή να επιφέρει σε σχέση με τον κανονισμό Ρώμη 1. Ε, στο ισχύον δίκαιο ισχύει Ε, ισχύουν τα εθνικά νομικά συστήματα. Δεν έχει νόημα να γίνουν συστάσεις στο πλαίσιο αυτό εφόσον δεν έχει τεθεί σε ισχύ το νομικό πλαίσιο το οποίο είχε σαν σκοπό να ε, πατάξει όλες τις ε, παραβιάσεις του ισχύοντος πλαισίου. Χωρίς μελέτη αντικτύπου αυτής της οδηγίας το να προτείνεται μια πολύ ευρύτερη οδηγία δεν έχει κανένα νόημα. Επίσης δεν υπάρχει δικαιολογία προκειμένου να περιοριστεί ο βασικό, η βασική αρχή της ελευθερίας των υπηρεσιών. Για παράδειγμα ο περιορισμός της απόσπασης για τη διάρκεια, σε μια διάρκεια 24 μηνών για ορισμένους κλάδους δεν έχει απολύτως κανένα νόημα και για κλάδους όπου πραγματικά υπάρχει τεράστιο αριθμό αποσπασμένων εργαζόμενων. Και θα ήθελα να πω ότι η εξισορρόπηση των αμοιβών στις χώρες μέλη δεν μπορεί να γίνει με την επιβολή ορισμένων ε, κανόνων. Πρόκειται για μια οικονομική διαδικασία η οποία θα έπρεπε να γίνει με έναν ε, φυσικό τρόπο. Εάν προσπαθήσουμε να το κάνουμε τεχνητά, αυτό θα είναι εις βάρος των επιχειρήσεων καθώς και των ε, καταναλωτών και των εργαζομένων. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα χάος που θα είναι εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων οι οποίες θα αναγκαστούν να μετατοπίσουν τις δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας ε, παράνομης ε, επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κάτι το οποίο είναι παράλογο. Ευχαριστώ κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δουλειά που έχει γίνει στην Επιτροπή Απασχόλησης. Συμφωνώ ότι αυτή η διαδικασία της κεντρική κάρτας δεν είναι πιστική Νομίζω ότι η Κομισιόν έχει δίκιο που παρουσιάζει την πρόταση αυτή και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος για να εγγυηθούμε παρόμοιες συνθήκες εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι η νέα πρόταση της Λογικής Προεδρίας για την εφαρμογή της έννοιας της ε, αμοιβής ε, για αποσπάσεις που είναι άνω των 9 μηνών, ενώ αυτές που είναι κάτω από 9 μήνες θα παραμείνουν ε, εντός της έννοιας των ελάχιστων ορίων μισθού. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα πραγματικό θέμα διάκρισης και διαφορετικής μεταχείρισης για παρόμοιες συνθήκες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου C396 κάθετος 13 είναι η υπόθεση των Φιλανδών ε, εργαζομένων που εργάζονταν στην εταιρεία ηλεκτρισμού και ουσιαστικά εκεί είχε εφαρμοστεί τη λέξη όρια μισθού για να καλυφθούν όλες οι αμοιβέ. Από ό,τι καταλαβαίνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για αυτή την υπόθεση. Έτσι λοιπόν, συνολικά, η πρόταση της Σλοβακής Προεδρίας όχι μόνο θα αποδυνάμωνε την εφαρμογή, αλλά ουσιαστικά θα παρέκλεινε και από την ερμηνεία του δικαστηρίου που οι κανόνες ε, της αμοιβή για τους ε, τοπικούς εργαζομένους ε, που προκύπτουν από συλλογικές συμβάσεις εφαρμόζονται επίσης και στους αποσπασμένου εργαζόμενου. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και να δούμε και τι ακριβώ συμβαίνει στο Συμβούλιο. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή οδηγία για τους αποσπασμένου εργαζόμενου. Είμαι επί της αρχής εχθρικό, γιατί αν και θέλει να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των αποσπασμένων εργαζομένων και των τόπιων εργαζομένων. Αντιθέτως, διατηρεί τη διαφορά του κοινωνικού άχθος γιατί θα συνεχίζει να πληρώνει ο εργοδότης το κοινωνικό άχθος της χώρα προέλευσης. είναι μια πρόταση που θέτει και θέμα επικουρικότητα ε, και ουσιαστικά αυτή τη λέγεται από την κίτρινη κάρτα που έχει κατατεθεί από 11 κράτη. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, παραβιάζεται συνεχώς. Καθώς είμαστε και στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είμαι απολύτω βέβαιο ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση. Θα σα την έκθεση Τβέλτ που ψηφίστηκε από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και προβλέπει ένα μηχανισμό αξιολόγηση στο βαθμό που να ξέρουμε ένα κράτο παραβιάζει το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Φυσικά αναφέρομαι στο μηχανισμό που προβλέπεται από το άρθρο 7 τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξέρετε ότι αυτή η πρόταση είναι σε αντίφαση κατάφορη με γνωμοδότηση της υπηρεσία, αστυνομική υπηρεσία του Συμβουλίου, που ερμηνεύει το άρθρο 7 και λέει ότι πρόκειται για μια διαδικασία εποπτείας που δεν περιλαμβάνει πρώτερη αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν δεν μας δίνει καμία νομική βάση. Έτσι λοιπόν αυτή η πρώτερη φάση αξιολόγησης που τίθεται όμως σε εφαρμογή από την έκθεση Ιντβελτ να δημιουργηθεί. Τι θα κάνει τώρα η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σα το ρωτώ, γιατί το πρόβλημα τη έκθεση Ιντβελτ είναι ότι δίνει αρμοδιότητα στην Κομισιόν να υιοθετήσει ένα πίνακα πορεία και συστάσεων και προσθέτει στο άρθρο 7 διατάξει που δεν θα έπρεπε να προσθεθούν. Έτσι λοιπόν, ρωτώ τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και πραγματικά σας δίνω την ευκαιρία να αποδείξετε ότι θέλετε να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας. Κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στην έκθεση του κυρίου Καβαντά για να σας πω ότι η ομάδα μας είναι ευνοϊκή προς την ε, πρόταση της Επιτροπής και ειλικρινά η αρχή ότι χρειάζεται ίση αμοιβή για την ίδια εργασία στον ίδιο χώρο ε, είναι θεωρώ θεμελιώδης αρχή που δεν μπορώ παρά να υπαρασπιστώ εντός ε, μιας Ευρώπη, Ευρώπης που ακριβώς μεριμνά για τον πολίτη. Και πιστεύω ότι εφόσον πρόκειται εδώ για ένα πρόβλημα διασυνοριακής φύσης δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να παραβιάσουμε την αρχή ε, της επικουρικότητας. Γιατί από τα δικαιώματα των χωρών μελών για να νομοθετήσουν και να διατυπώσουν τις ε, προϋποθέσεις εργασίας. Άρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταλάβω αυτό, αυτή την ένσταση που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας και χαιρετίζω την προσπάθεια της ε, Επιτροπής να εξετάσει τι ε, τις κίτρινες ε, κάρτες. Κύριε Πρόεδρε, κατάλαβα σωστά ότι αποστήλατε μια επιστολή προς την νομική υπηρεσία με, που περιλαμβάνει πολλά ερωτήματα. Ε, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα αυτά. Απλώ θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι για το γεγονό ότι ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση και συμφωνώ με το χρονοδιάγραμμα. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω παρόλα αυτά εδώ ότι ο σκοπό τη ενία αγορά είναι να δημιουργηθεί ένας ενάρετος οικονομικός ε, ε, κύκλος και όχι να γίνει κοινωνικό dumping και να υπονομευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια βασική αρχή, η οποία θα έπρεπε να μας καθοδηγεί στις μελλοντικέ μας πράξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πω κάποια πράγματα ο κύριος Χρυσόγονος θέλει να πάρει το λόγο. Επιτρέψατε μου να κάνω κάποια σχόλια. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας εδώ, γιατί μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό θέμα το οποίο θα πρέπει να το προσεγγίσουμε με ενιαίους ε, κανόνες και θα πρέπει πραγματικά να καλύψουμε τα ελλείμματα και να διορθώσουμε τα διέξοδα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία λοιπόν. Εγώ θα κάνω μια παρέμβαση στα τσεχικά, στα για να είμαι πιο ακριβής. Σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής θεωρώ ότι δεν είναι ισορροπημένη. Ε, και, κυρίως όσον αφορά, αφορά θέματα της εσωτερικής αγοράς. Η έλλειψη ισορροπίας σημαίνει ότι από τη μία εξετάζονται μόνον θέματα αποδοχών και όχι ουσίας. Από την άλλη, αφαιρεί από τις επιχειρήσεις των νέων χωρών μελών το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο είχαν και το οποίο συνεχίζουν να έχουν στην πραγματικότητα. Όσον αφορά τις ακραία κινητικές επιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις στον, τομέα των ε, μεταφορών, για παράδειγμα, ε, δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στο πλαίσιο αυτής της πρότασης. Υπάρχει ένα μέγιστο όριο για την διάρκεια της περίοδου απόσπασης, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια ελάχιστη διάρκεια. Για την οποία να ισχύουν αρχές όπως ίση αμοιβή για την ίση εργασία. Ε, θα πρέπει να συζητήσουμε αρχές όπως ε, ίδια αποδοχή, ε, ίση αμοιβή για το ίσο έργο, για την ίση εργασία εντός μιας επιχείρησης όταν μιλάμε για μια ενιαία εσωτερική αργόρα. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να πληρώνεται διαφορετικά ένας υπάλληλος της ίδιας εταιρεία στη Γερμανία από έναν υπάλληλο της επιχείρησης αυτής στην Τσεχία. Υπάρχει ένας τοξικός χαρακτήρας αυτή την ε, πρόταση γιατί ορισμένες επιχειρήσεις, ορισμένα μέρη της Ευρώπης όπως σας είπα θα απολέσουν το συγκριτικό τους ε, πλεονέκτημα. Και τότε θα ανακύψει το ερώτημα κατά πόσο επιχειρείς από τις, ε, τα παλαιότερα μέλη ε, δεν θα χάσουν τα, ε, δεν θα πρέπει να χάσουν τα πλεονεκτήματα τα οποία είχαν στην πρώτη περίοδο της εισδοχής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για μια συζήτηση που συνεχίζεται μετά και την εξέταση των ε, κειμένων ε, που έχουν εξετάσει οι επιτροπές μας. Ε, σας υπενθυμίζω την περίφημη οδηγία Μπόλκενστάιν και άλλες, όπου είχαμε τεράστιες αντιδράσεις, κάποιες φορές και δικαιολογημένα. Βεβαίω, όλε αυτέ οι διαμαρτυρίε συνήθω σε εθνικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια τη εθνική εκλογική εκστρατεία, ε, έλαβαν χώρα. Τώρα, αν αυτό το νέο κείμενο θα είναι μια πανάκια που θα λύσει όλα τα προβλήματα, όχι, ούτε εγώ το πιστεύω. Όμω, θα ήθελα να σα πω δύο πράγματα. Οι νόμοι γίνονται για να υπηρετούν τις αρχές, όχι το αντίθετο. Δεν ε, ε υπονομεύονται οι αρχές ε, για να επικρατήσει το δίκαιο. Οι νόμοι υιοθετούνται λοιπόν για να εξυπηρετούν τις αρχές. Ποιες είναι οι αρχές που εδώ πέρα θεωρούμε πιο σημαντικές. Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όντως πετύχει την ελεύθερη κυκλοφορία των ανδρών και γυναικών, κεφαλαίων, επενδύσεων Το χρήμα λοιπόν, το οποίο δημιουργεί πλούτο, έχει οργανωθεί και δομηθεί με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζετε κι εσείς όμως ότι η δημιουργία πλούτου έχει δύο σκέλη και όχι ένα. Είναι και το κεφάλαιο, το χρήμα, αλλά είναι και το μισθολογικό κεφάλαιο ή μάλλον ανθρώπινο δυναμικό. όπως λέει και ο Μαξ, ε, τον οποίο δεν στηρίζω, αλλά ε, τον έχω διαβάσει επισταμένος και έτσι γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτόν. Αναφέρεται λοιπόν ότι η Επιτροπή ε, ε, θέλει να αντιμετωπίσει μία κατάφορη αδικία και συνεχώς κατακρίνεται αυτή η αδικία με βάση ότι η σημερινή κατάσταση των αποσπασμένων εργαζομένων οδηγεί στην καταστροφή επιχειρήσεων, το οποίο ισχύει, στην πανατόπιση με την κατάσταση των επιχειρήσεων, και αυτό ισχύει, ή ότι έχουμε και αυτή την παράνομη ή ανήθικη ε, πρακτική ε, των ε, επιχειρήσεων ταχυδρομικής θηρίδας για λόγους φοροδιαφυγής ουσιαστικά. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια με κάποιον τρόπο εάν η Επιτροπή δεν αντιμετωπίσει παρά μόνο την ισοδύναμη αμοιβή από όπου και αν βγαίνουν, από και αν έρχονται αυτοί οι εργαζόμενοι, Κανείς δεν πρέπει να πει κάτι ενάντια σε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας ε, Βούλγαρος ε, υπήκος να αμείβεται στη Γαλλία λιγότερο από τον Γάλλο, για παράδειγμα. Επομένως, ευσταθούν οι κριτικές, αν και ακούμε μόνο κριτικές. Τώρα μπορούμε να θίξουμε το ζήτημα της ε, κοινωνικής προστασίας και της χρηματοδότησής της. Ένας εργαζόμενος από την Πολωνία, όπως αναφέρεται πολύ στις, δυστυχώς στις εκλογικές εκστρατείες. ορθώς θα παίρνει τον ίδιο ε, μισθό αν εργάζεται στη Μεγάλη Βρετανία. Εντάξει, τώρα πλέον η Μεγάλη Βρετανία θα μας απασχολεί. Ε, ή στην Ιταλία να παίρνει τα ίδια με έναν Ιταλό. Ναι. Όλα τα κοινωνικά κινήματα το απαιτούν. Και αντικειμενικά μας σας πω, εντάξει λυπάμαι, αλλά οι Πολωνοί, οι Βούλγαροι, οι Τσέχοι οι εργαζόμενοι με τα χαράς λαμβάνουν έναν καλύτερο μισθό ε, σε μια χώρα που μπορούν να πάρουν καλύτερο μισθό, γιατί ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Προσπαθούν να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα πράγματα, να τα μαζέψουν, για να χτίσουν κάτι όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Και αν σεβο... θέλουμε να σεβόμαστε τους ανθρώπους, πρέπει να τους δίνουμε ίσα δικαιώματα από όπου και αν προέρχονται και τέτοιες εγγύησεις. Βεβαίως, συμφωνώ με αυτό που ανέφερε ο Πρόεδρος, δεν είναι πλήρως το κείμενο. Γιατί πράγματι οι κοινωνικές ε, παροχές θα είναι λιγότερες ανάλογα με τον μισθό για ένα άτομο το οποίο ε, είναι εργαζόμενο σε απόσπαση. Γιατί δεν θα έχει και, τη... και την ίδια κοινωνική ασφάλιση, τις ίδιες εισφορές ε, ένας Πολωνός, για παράδειγμα, εργαζόμενος με τον Γάλλο ή τον Ιταλό ναι, όντω θα πρέπει κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Αλλά ε, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αυτό το βήμα, το οποίο ακυρώνει μία από τις πιο σημαντικές ε, στρεβλώσεις και έχουν καταγγείλει πολλές φορές ε, πολλά κόμματα, ακόμα και τα ακραία κόμματα κάποιες φορές. Το κάνουμε λοιπόν αυτό το πρώτο βήμα, γιατί είναι στο πεδίο βολής μας και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Επίσης, εάν οι κοινωνικές εισφορές στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εργαζόμενοι είναι πιο χαμηλές και αυτό συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένα Πολωνό εργαζόμενο που έρχεται στη Γαλλία, αν έχει τον ίδιο μισθό με έναν Γάλλο εργαζόμενο, το οποίο είναι καλό, και πάλι ε, σε μία ώρα θα είναι διαφορετική η αμοιβή του, γιατί οι εισφορέ που πληρώνει ένα Γάλλο για την ασφάλιση τη εξαιρετότητα κτλ. είναι πολύ πιο σημαντικέ. Παραμένει λοιπόν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Φαντάζομαι το έχει σκεφτεί η Επιτροπή και μάλλον γι' αυτό το λόγο ε, επιλέγει να εξετάσει ένα θέμα τη φορά. Από τα ακραία κόμματα έχω ακούσει και πάλι κάποιες φορές ευσταθούν τα επιχειρήματα για την μετεκατάσταση των επιχειρήσεων. Όμως πρέπει να χαιρετήσουμε αυτό το βήμα που γίνεται προς τα μπρος. Λυπάμαι αν σας στεναχωρώ, σας ενοχλώ ή σας σοκάρω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος της εξέτασης του σημείου 7. Περνάμε στο σημείο 8. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την παραβίαση των δικαιωμάτων γενοδιτικής ιδιοκτησίας ο κύριος Καβαντά και ο κύριος Βεύκα στη συνέχεια. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. E, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Καβαντά και ο κύριος Ράπκα μετέβησαν στο Αλκάντε για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Και υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρχε και αρκετές με κυβερνητικές οργανώσεις που συνεργάζονται με την κυβέρνηση του Λικάντη για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής δικτυσίας. Ο Ζαν Μαρκαβαντά ήταν ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας εγώ για πρώτη φορά παρευρέθηκα σε μια τέτοια συνάντηση. Για μένα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κυρίως ε, όταν άκουσα τις διάφορες ε, απόψεις και τους διάφορους ε, τρόπους χρήσης των μοντέρνων τεχνολογιών, αλλά και ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τι έχουν να πούν οι εκπρόσωποι μας που εργάζονται στο Αλκάντε, στον οργανισμό του Αλκάντε. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι μέρες και ελπίζω ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ αυτής της Επιτροπής ε, και του Agency στο Αλκάντε. Ένα σημαντικό μέρος Τη ε, σχετική νομοθεσία θα περάσει από τη δική μα επιτροπή. Έτσι λοιπόν ε, είναι απαραίτητη η συνεργασία με τον οργανισμό στο Αλικάντε. Ο Ζων Μαρή από την πλευρά του θα παρουσιάσει κάποιε πιο λεπτομερεί πληροφορίε. Δεν θα ακρηγορήσω. Θα συμφωνήσω, μα είπε ο κ. Ζιέφκα, αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή σα στο εξή. Πρόκειται για έναν οργανισμό που δεν είναι γραφειοκρατικός, ε, ούτε έχει υπερβολικά πολλούς υπαλλήλου, χρησιμοποιεί τους πόρους με πολύ αποτελεσματικότητα και τρίτον ε, πρέπει να διατηρήσει και την ελευθερία διαχείρισης και οργάνωσης αυτός ο οργανισμός. Γιατί εγώ υποψιάζομαι ότι κάποιος ε, θέλει να καταστήσει πιο πολύπλοκο τον καθεστώς λειτουργίας αυτού του οργανισμού Ε, τώρα, ε, αν θα μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση και πιο αποτελεσματική, πρέπει να το δούμε στα πλαίσια τη επικουρικότητα. Πρόκειται για έναν οργανισμό που πηγαίνει πολύ καλά και πρέπει να τον αφήσουμε να εργάζεται στην ησυχία του. Ανήκει ε, στο γραφείο παρακολούθηση τη νέα αγορά, τη εσωτερική αγορά τα καθήκοντά της ε, είναι να παρατηρεί αν ε, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα διανοητικής διεκτησίας ε, και ξέρετε οι μεγάλες επιχειρήσεις πολύ εύκολα μπορούν να περισπιστούν τον εαυτό τους όμως οι μικρές επιχειρήσεις στρέφονται προς το παρατηρητήριο για να τις βοηθήσει. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει τις ε, πληροφορίες που αφορούν τους οργανισμούς που λειτουργούν καλά, να τις διαβιβάσουμε και στο κατάλληλο επίπεδο. Ήθελα απλώ να πω ότι έκανα μία πρόταση και έθεσα το θέμα στην Ολομέλεια της αναγκαιότητας να εξηγήσουμε τι συμβαίνει με τη βιομηχανία της παραποίησης. Πρόκειται για τεράστια παγκόσμια βιομηχανία και φυσικά δεν πλουτίζουν μόνο όσοι παραποιούν. Και για μια ακόμη φορά πρέπει να θεωρήσουμε ότι ακόμη και αν πρέπει να σεβαστούμε την επικουρικότητα, πρέπει να δούμε και την διασυνοριακή πτυχή αυτού του εγκλήματος. Ε, ουσιαστικά πρόκειται για μια κούρσα που δεν τελειώνει. Όσο περισσότεροι παραποιητές ε, υπάρχουν, τόσο πιο πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τον οικονομικό ιστό μας. Αυτό το θέμα συστήθηκε πάρα πολύ θετικά και θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά επικεντρωθήκαμε στο ότι θα πρέπει να στραφούμε προς μια νομοθεσία πολύ πιο δεσμευτική απέναντι στο φαινόμενο της ε, παραποίησης και η απάντηση στις ερωτήσεις που τέθηκαν ε, ήταν ε, ότι δεν ναι, πρέπει να ενισχύσουμε πάρα πολύ τα μέσα παρατήρησης και τα μέσα καταστολής. Αυτό περνά από μία υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών και ουσιαστικά εδώ εμπλέκονται και πολλές εισαγγελίε και για να μην πω και η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία. Τελικά δεν ε, πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι ο καθένας μπορεί να δυσδεί με οποιοδήποτε τρόπο θέλει σε αυτή την αγορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 26. Ε, ε, ανταλλαγή απόψε για ένα μηχανισμό που εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την ε, ειρήνη. Si j'avais su, je serais venu plus αν το ήξερα θα είχα έρθει πιο αργά. <laughs> Λέει ο κύριος Καβαντά. Η έκθεση αυτή για τη νομική βάση του κανονισμού για ένα εργαλείο που να συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο ε, μιας ψηφοφορίας σήμερα. Ε, γιατί πραγματικά έχουμε συζητήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό στις προηγούμενες συνεδριάσεις μας. Παρ' όλα αυτά, ε, οι σοσιαλιστές ε, θέλουν να ζητήσουν την αναβολή της ψηφοφορίας έως ότου η ΑΦΕΤ, η οποία νομοθετεί επί της ουσίας, να μπορεί να τοποθετηθεί εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο είστε σύμφωνοι. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην περίπτωση αυτή ε, θα πρέπει να πείτε κατά πόσο επιθυμείτε να συνεχίσω εγώ να είμαι εισηγητής ε, στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και εφόσον ο πρόεδρος μου το επιτρέπει θα δώσω το λόγο στις ε, πολιτικές, ε, θα δοθεί ο λόγος στις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Φως έχει καταρχήν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ε, ευχαρίστως είμαστε διατεθειμένοι να ξεκονομηθεί ο χρόνος Όχι, να, μην, να, να δοθεί ο χρόνος εφόσον μια άλλη ομάδα επιθυμεί να συζητηθεί το θέμα. Εγώ... Ε, And I will ε, Θα μιλήσω, θα διαβάσω τη δήλωση της συναδέλφου, η οποία γέννησε το παιδί της και δεν μπόρεσε να παραστεί. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδες που συμφώνησαν να αναβληθεί η ψηφοφορία για τη νομική βάση όσον αφορά την πρόταση της εκπόνησης ενός νέου εργαλείου που να συμβάλλει σταθερότητα και στην ειρήνη. Στη βάση των διαφόρων απόψεων τα οποία παρουσιάστηκαν στη Γιούρη ε, στο παρελθόν πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δούμε τα διαφορετικά επιχειρήματα και να τα σταθμίσουμε πριν προχωρήσουμε στη ψηφοφορία για την νομική βάση. Γιατί από τη μία ε, υπάρχει αναμφίβολα η ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη συμβολή της για την υποστήριξη της διαδικασίας ειρήνης και σταθερότητας σε ένα ευάλωτο πλαίσιο, ιδιαίτερα όταν δούμε τις ε, ταχείες αλλαγές σε θέματα ασφαλείας. Από την άλλη είναι σημαντικό το νέο εργαλείο για τη σταθερότητα και την ειρήνη να θεσπιστεί ε, σε ευθυγράμμιση ε, με τους άλλους ε, βιώσιμους αναπτυξικούς στόχους, ούτω ώστε να είναι αποτελεσματικό και να συμβάλλει πραγματικά σε μια βιώσιμη ειρήνη. Εάν οι προταθήσεις δραστηριότητες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν ε, από το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι ε, με τα κριτήρια της αναπτυξιακής ε, βοήθειας που έχουν αποφασιστεί από κοινού με τον ΩΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι η, η κατάρτιση για το στρατό μπορεί να είναι επιλέξιμη μόνο σε ζώνες όπου δεν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή η προταθήσα νομική βάση για την ανάπτυξη και τη συνεργασία, άρθρα 2, 1, 9 και 12 δεν ισχύουν. Η κατάρτιση του προσωπικού Όσον αφορά την κατάρτιση προσωπικού και τι άλλε υπηρεσίε, η Γραμματεία δεν επιτρέπει τον εφοδιασμό εξοπλισμού που θεωρείται ε, ως εξοπλισμός ο οποίος ε, χορηγείται σε μία χώρα εταίρο. Ε, η πρόταση δεν περιορίζεται στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας. Η ομάδα μας θεωρεί λοιπόν ότι είναι πιο λογικό να αναμένουμε τα αποτελέσματα της ε, ε, έκβασης των διαπραγματεύσεων στις άλλες επιτροπές ε, ανάπτυξη, για παράδειγμα, πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για τη νομική βάση. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι θυμάμαι ότι θέλαμε να περιμένουμε την νομική σύσταση του Συμβουλίου δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν κάποια νέα από εδώ. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ για να καταλάβω πόσο ακριβώς θα χειριστούμε αυτό το θέμα σήμερα. Να πω και εγώ δύο λόγια λοιπόν. Παρότι στηρίζω το αίτημα των σοσιαλιστών για αναβολή της ψηφοφορίας, επιτρέψτε μου λοιπόν ε, να εκφράσω την ισχυρή μου έκπληξη όταν διάβασα την απάντηση της Επιτροπής στο έγγραφό μας. Είχαμε ζητήσει από τη θυμάστε, από την νομική υπηρεσία ή μάλλον από την Επιτροπή να μας ε, δώσει τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της. Ο Λουίς Ρομέρο Ρικουέρα απέστειλε λοιπόν επιστολή σε αυτή την Επιτροπή, την οποία έχουμε λάβει τουλάχιστον ως συντονιστές και στο βράδυ, με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου και ισχυρίζεται ότι η νομική υπηρεσία τη Επιτροπή δεν έχει συντάξει γνωμοδότηση όπου θεωρεί ότι η νομική βάση τη πρόταση ε, της οικοδόμηση δυναμικού ε, την χάνει επεξεργασία. Έχω, είμαι έκπληκτη γιατί έχω ακόμα και τον αριθμό καταχώρηση αυτού του εγγράφου. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολουθεί τις ε, αρχής της ε, καλή την πίστη ε, συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και θα πρέπει να αναλυθούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Προτείνω λοιπόν στην τεμία να επαναλάβουμε το αίτημά μα για αυτό το έγγραφο με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν. Ιδάλω είναι αδύνατο να συνεχίσουμε την εξέταση αυτού του ζητήματο στην Επιτροπή μας. Και νομίζω ότι η κυρία Ντελβό πολύ σωστά λέει ότι έχουμε ζητήσει και από το Συμβούλιο ε, ε, γνωμοδότηση τη νομική Υπηρεσία. Βέβαια αυτή η συζήτηση δεν έχει να κάνει με τη διασύνδεση ασφάλεια και ανάπτυξη. Εξετάζουμε τη νομική βάση. Όπω και να έχει, νομίζω ότι ε, νομοθετικά μέτρα θα πρέπει να βασίζονται σε κατάλληλη νομική βάση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συνεχίσουμε ε, επιμελώς να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα. Κύριε Χρυσόγονος. Κύριος Χρυσόγονος. Wait a minute. Περιμένετε ένα λεπτό. Κάτι περίεργο έχει διατύπωση στην επιστολή που σας απευθύνεται από τον κύριο Λουίς Ρομέιρο Ροκέινα. Λέει, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχει καμία γραπτή γνωμοδότηση. <laughs> What is happening? Yeah. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς. So, ε, native speaker says that should is correct. Οι φυσικοί ομιλητές βέβαια λένε ότι, το should εδώ είναι σωστό. Δεν ξέρω αν κάποιος από την Επιτροπή θέλει να σχολιάσει. Όχι μάλλον. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε την πρόταση της κυρίας Χάουταλα και να επαναλάβουμε το αίτημά μας. Ο κύριος Καβαντά. Όχι, κανείς δεν θέλει να πάρει το λόγο. Έχετε δίκιο. Θέλω να διευκρινίσω ότι η Επιτροπή έγραψε σαν έπρεπε να καταγραφεί το γεγονός ότι δεν θα υπήρχε γνωμοδότηση. Το σκέφτηκε, αλλά δεν Δεν υπάρχει γνωμοδότηση και το Συμβούλιο δεν έχει απαντήσει. Δεν έχουμε λάβει τίποτα από το Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, ε, νομίζω ότι σωστά είναι τα όσα είπε η κυρία Ντελβο και Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εξαντλήσει και αυτό το σημείο. Και θα συνεχίσουμε με τις συνεδρίες των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Όποιος λοιπόν δεν έχει δικαιωμένα βρίσκεται στη συνεδρίες και κλεισμένων των θυρών, την αίθουσα.